Take a seat. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε. Good morning. Good morning. Möchte Sie herzlich an diesem frühen Morgen begrüßen. Darf Sie bitten, die... Λοιπόν, σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά. Σας καλημερίζω θα ήθελα να σας μεταφέρω τις αποφάσεις των συντονιστών που έγιναν χθε δεκτές. Αν δεν συμφωνείτε μέχρι τις 12 μπορείτε να εκφράσετε τη διαφωνία σας. Ε, μπορείτε να πάρετε τις κάρτες σας όμως για να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσουμε με την πολιτιστική διάσταση της εξωτερικής δράσης. Η κυρία Σάκε. Ευχαριστώ Ντόρις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την επικοδομητική τους συνεργασία. Νομίζω ότι στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Πρόκειται για θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το δυναμικό το οποίο έχει στη διάθεσή της στον τομέα του πολιτισμού. Καλώς, ξεκινάμε λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Όχι, συγγνώμη, συμβιβαστική Ένα Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 43 λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 48 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 49 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κοιτάξτε θα μείνω στα αγγλικά να μην σας μπερδεύω. Αυτά τα αγγλικά είναι επαρκή λοιπόν. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία της εισηγήτριας 2 υπέρ κατά αποχές. Πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινάμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Λοιπόν, θα ξαναρχίσουμε την ψηφοφορία πάνω στην δεύτερη, την προφορική υπαριθμών 2, λοιπόν, της εισηγήτριας. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκατέσσερις υπέρ, δέκα κατά. Δεκαπέντε υπέρ λοιπόν και 10 κατά δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 77 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 79 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 79 ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Λοιπόν, 13 υπέρ, 10 κατά δεκτή. 80 υπέρ, κατά. Αποχές, δεκτή. 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή 83 υπέρ συγγνώμη 87 υπέρ κατά αποχές απο, απορρίπτεται ή μάλλον ηλεκτρονικός έλεγχος για την 87 τέλος 17 κατά, 8 υπέρ απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 101 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 98 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 102 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 100 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή 115 και 116 ταυτόσημοι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 115 Τέλος. 20 υπέρ 6 κατά. Δεκτή λοιπόν. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 123 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 123 Τέλος. 11 υπέρ, 14 κατά απορρίπτεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο 11 υπέρ, υπέρ ψήφισε η Κώστα, 20 υπέρ, 14 κατά. Απορρίπτεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 126 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 127 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 128 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 129 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 130 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. Δεκτή είπαμε. Οκ, okay, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 137. Τέλος. 15 υπέρ, 13 κατά. Συγγνώμη αν βιάστηκα, αλλά 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ή μάλλον ηλεκτρονικός έλεγχος για την 139. Τέλος. 15 κατά και 11 υπέρ. Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 141 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45-46 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές 147 150 μάλλον, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 151 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 151. Τέλος της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 9 κατά. 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά 153 ναι, υπέρ, κατά. Δεκτή λοιπόν. 154 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 160 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 161 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, ή μάλλον έλεγχος για την 161. Τέλος του ελέγχου. 15 υπέρ 13 κατά δεκτή. 163 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 166 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 166. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 13 υπέρ 13 κατά. Θέλετε κάτι να προσθέσετε. Εγώ απλά εφαρμόζω τους κανόνες, δεν αποφασίζω. Εκατόν εξήντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 167 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Προφορική 4, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές δεκτή 171 υπέρ κατά αποχές Λοιπόν, 171 υπέρ. Αλλάξατε γνώμη. Ίσως πάω πολύ γρήγορα. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 176 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 178 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική ή 179 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 183 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 188 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 188. Τέλος. 19 υπέρ, 7 κατά δεκτή. 189 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 14 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ, κατά αποχές δεν είναι ξεκάθαρο, ψηφίζουμε την 13. Τέλος. 17 υπέρ 10 κατά. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές Για την 24 ξαναψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. 9 ε, ναι, υπέρ 18 κατά. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ όχι. 28-28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 33 και 34 υπέρ κατά αποχές δεκτές 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 35 μου άλλαξαν την κάρτα και δουλεύει πλέον λέει Κώστα πέρα στις ψηφοφορίες 15 υπέρ 12 κατά γίνεται δεκτή. Mm. 19, συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή τρία υπέρ κατά αποχές απο, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τρία. τέλος δεκτή Τοπολογία 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 5 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 7 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 9 υπέρ, κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 9. Τέλος. Απερίφθη. Λοιπόν, τελική ψήφος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 26 υπέρ, 0 κατά, συγχαρητήρια. Είναι η πρώτη φορά που ψηφίσατε μαζί μας. Not you. No. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να πείτε κάτι, όχι, εντάξει. Ο oh, Μαράκη, everything is okay, εντάξει, εντάξει. Μαράκη, μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία. Λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, δύσκολο η κυρία Μαρίτα Σμιτ. Θέλετε να πείτε κάτι κυρία Σάντσε Σμιτ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι βελτίωσαν με τις τροπολογίες τους και τις εξαιρετικέ τους ιδέες. Θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη ε, σχετικά με αυτές τις βιομηχανίες που παρουσιάζουν ένα τεράστιο ενδιαφέρον για την οικονομία μας. Ελπίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις εφάνταστες δραστηριότητες. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει να εξελιχθεί σωστά η οικονομία μας. Ευχαριστώ. Και εγώ λέει η κυρία Πακ στα γαλλικά θέλω να ευχαριστήσω την γραμματεία γιατί ακόμα και χθε τη νύχτα μας έστειλαν την τελική, τον τελικό κατάλογο ψηφοφορίας και η κυρία Κώστα θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για την ε, δεκτικότητά της. Εγώ σας και η εισηγήτρια της σοσιαλιστικής ομάδας συνεισφέραμε, ε, δώσαμε πολλά στοιχεία δικά μας, τα δέχτηκε η εισηγήτρια και την ευχαριστώ επίσης και για την αποδοχή της δημιουργίας ενός λευκού βιβλίου για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ και τη γραμματεία επίσης γιατί έκανε τεράστια προσπάθεια σε ένα δύσκολο θέμα. Εσείς όχι, εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσω γερμανικά πια. Υπέρ κατά αποχές. Εντάξει, απλά πράγματα. Υπέρ κατά αποχές. Für dagegen Μπορούμε να τα πούμε και ελληνικά. Κατά. Ακούγεται ωραία. Πολύ καλά. Ξεκινάμε λοιπόν. Τροπολογία 52. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 53 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας λοιπόν αποτέλεσμα απορρίφθηκε 13, 13 υπέρ 15 εναντίον 54 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Ρέγγι 11 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 11 της Ρέγγι άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας 17 εναντίον 10 υπέρ απορρίφθηκε Ήτρε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 59 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 60 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 68 σε τμήματα ψήφιση πρώτο τμήμα υπέρ κατά Α, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της 68 ε, πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα 15-14 εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε πάλι ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα τη 68. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία Αποτέλεσμα. 16 εναντίον 13 υπέρ απορρίφθηκε. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή 75 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 76 υπέρ κατά α... τι είπατε να ελέγξουμε λέτε ηλεκτρονικά Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 75 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 18 εναντίον 11 υπέρ. Δεν μπορεί να πάει χειρότερα. Καταψηφίστηκε. Λοιπόν. Εντάξει, που είχαμε μείνει. 76 τώρα υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 138 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε την 138 πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα 20 υπέρ 9 εναντίον εγκρίθηκε μάλιστα Απασχόληση 22 υπέρ όχι συγγνώμη 78 λέτε εντάξει εκεί κάτω συγγνώμη ναι Ωραία, 78. Σε δύο τμήματα λοιπόν. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Προφορική τροποποίηση. Σίλβια Κώστα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 82 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Να ρωτήσω κάτι. Λόκεγκαρτ. Χθες είχατε αναγγείλει ότι πρόκειται για μια τροπολογία. Την έχετε. Θέλετε να την αναφέρετε. Τι γίνεται. Χθε σα το είχα πει, ότι πρέπει σήμερα να μας το πείτε, γιατί θα ψηφιστεί σήμερα. Τι γίνεται. Κυρία Σάντσες, τι λέτε. Όχι. Εντάξει, τότε συγγνώμη. Ωραία. Έτσι νοιάζομαι εγώ για τους φιλελευθέρους, φίλε μου. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιος με ευχαριστεί γι' αυτό, κανείς. 84 υπέρ. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 84. Τέλος ψηφοφορίας. 23 εναντίον. Απορρίφθηκε. Λοιπόν, πάει αυτή. 86 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 87 υπέρ. Τι λέτε. 85 πρωτά. συγγνώμη, 85, σωστό, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε 87 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε προφορική τροποποίηση 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 89 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε της απασχόλησης 16 υπέρ, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 92 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 94 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 95 και 96 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 97 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 99 και 98 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 104 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 102 υπέρ κατά αποχές τι λέτε 102 η 102 δεν αποσύρθηκε. Η 102 δεν αποσύρθηκε. Λοιπόν και πάλι 102, 102 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 107 υπέρ κατά αποχές δεκτή 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 109 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 113 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 115 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 116 και 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 121 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 125 υπέρ κατά τι λέτε εσείς 125 δεν αποσύρθηκε η 125 είναι σαφές αυτό στα γερμανικά αυτό που είπα έτσι ξεκάθαρο φταίνε οι διερμηνείς λέτε ε δεν πειράζει 125 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Γιούρι 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 129 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Ήτρε 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 130 όχι τι λέτε καταπίπτει η 131 λοιπόν η 131 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 132 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 134 σε τρία τμήματα Ωραίο, επειδή είναι τόσο όμορφη. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. απόχέ απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. απόχέ απορρίφθηκε. Τρί... Κυρία Κώστα, για τη δική σας τροπολογία ψηφίζουμε. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. απόχέ απορρίφθηκε. Είδατε, αν συμμετείχατε θα ήταν άλλο το αποτέλεσμα. Τέλο πάντων, 136 υπέρ. υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίθηκε. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Έμπρο 23, απασχόληση 23, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 140, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 141, υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, έρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 141. Μάλιστα, 141. Πέρας ψηφοφορίας. Λοιπόν, 16 υπέρ, 13 εναντίον, υπεψηφίστηκε, εγκρίθηκε. 135 υπέρ. Τι λέτε εσείς, Ήτρε 10 λέτε, μάλιστα, συγγνώμη. Λοιπόν, πάει αυτή, Ήτρε 10 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 142, δεν θα ψηφιστεί λέει αυτή. 143 λοιπόν, υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε που πάμε 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 646 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 147, συγγνώμη 146 ήταν πριν, 147 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Έμπλο 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ρέγγι 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ρέγγι 8 υπέρ κατά κατά αποχές απορρίφθηκε. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 152 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε προφορική τροποποίηση 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 157 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 158 Α, πάει αυτή 159 160 τώρα υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 161 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 163 υπέρ κατά Αποχές. Θα ελέγξουμε. έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 163. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 15 υπέρ 14 εναντίον εγκρίθηκε. 166 υπέρ κατά αποχές. Εσείς είστε υπέρ, έτσι. Δική σας τοπολογία. Όχι. Α, συγγνώμη, λάθος μου. Λάθος μου, ζητώ συγγνώμη. 164 και πάλι. 164 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 165 αποσύρθηκε. 166 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 167 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 171 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 173 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 174 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε ήτρε 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 176 ε, υπέρ κατά και πάλι επαναλαμβάνουμε 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 177 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 178 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 179 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 181 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 15 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 19. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 18 εναντίον 11 υπέρ. Απορρίφθηκε 20. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε είναι 1 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την ίντα 1 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε την ίντα 1 πέρας ψηφοφορίας 15 εναντίον 14 υπέρ απορρίφθηκε 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε προφορική τροποποίηση 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή ήτρ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 30 όχι η 31 31 λοιπόν Κώστα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 32 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συνάδελφε Κέλλη τώρα τι είναι, βρίσκεται στην Ιρλανδία και πίνει υπέρ του Αγίου Πατρικίου. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ναι, μας το είχε πει. Πρέπει λέει να πάει στην Ιρλανδία να πει και ένα ποτηράκι. Δεν το επινόησα εγώ. 37 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε, ψηφίζουμε την 37 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. τι γίνεται εδώ. 20 εναντίον 9 υπέρ απορρίφθηκε. Εμπρ γάμα σι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε ρέγγι 1 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 42 υπέρ κατά και πάλι επαναλαμβάνουμε θα ελέγξουμε κιόλας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 κατά αποχές απορρίφθηκε η τρία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η επτά υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η οκτώ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η εννέα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και τώρα τι είναι, ίντερ είναι, τι λέει. Λοιπόν, μπορούμε να συμπτύξουμε μερικές τροπολογίες να τις πάρουμε ομού. Όχι, δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Ίντα, τι έχουμε εδώ. Είναι τα δύο. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Καταψηφίστηκε, απορρίφθηκε. Λοιπόν, τι είναι εδώ, πρόταση, suggestion. Λέω τώρα τους αριθμούς. Τρία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ερωτώ. 4, 5, 6, 7 μέχρι 9 μπορούμε να τις πάρουμε από κοινού, να ψηφίσουμε όλες. Γίνεται, τι λέτε. Όχι, τέλος πάντων. Πάντα κάτι ξεχωριστό. 4 υπέρ λοιπόν. 4. Αφού δεν επιθυμούν. Λοιπόν, τέλος πάντων. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 7 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 8 9 συγγνώμη υπέρ κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 9 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε την 9 πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα εγκρίθηκε βλέπετε εγκρίθηκε 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε έμπρο τώρα. Επιτροπή απασχόληση 1. Υπέρ κατά απορρίφθηκε. 2. Υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 3. Υπέρ κατά Αποχέ απορρίφθηκε. Να δεν θα ψηφιστεί, δεν θα ψηφιστεί η 6 τώρα. 6 υπέρ κατά απόχέ απορρίφθηκε. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 9 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 11 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η, 10, η 12 διορθώνει η υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 17 δεν θα ψηφιστεί. Η 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Η 19 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίθηκε. 20 υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίφθηκε. 21 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίθηκε. 24 υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίφθηκε. 25 υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίφθηκε. 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 28 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 30 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 31 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 32 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε ΑΒΓ τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκαν. Λοιπόν, πάει αυτό. Θεέ μου, τι γίνεται, είτε... Έβγαλε μαλλί γλώσσα μου. Λοιπόν, είτε τρία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Πέντε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Έξι υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε 7 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 8 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 9 και σε τμήματα κιόλα για όνομα του Θεού. Λοιπόν, 9 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 11 ε, δεν χρειάζεται να ψηφιστεί αυτή. Η 12 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 14 δεν θα ψηφιστεί ούτε η 15. Η 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Ρέγγι τώρα. 2 υπέρ Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 2 της Ρέγγι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε. Ρέγγι 2. Ψηφίζουμε. Ρέγγι 2. Βλέπετε. Μάλιστα. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 17 υπέρ 12 εναντίον εγκρίθηκε. Μα πώς πήγατε, πώς ψηφίσατε έτσι αντίθετα. Και πράσινη. Πρέπει να ακολουθείτε εσείς. Όχι εμένα. Το συντονιστή, το συντονιστή σας να ακολουθείτε εκεί. 17-12 εν πάση περιπτώσει εγκρίθηκε. Ποια ήταν οι δύο ήταν. Μάλιστα. Πάμε στην τρία. Τρία τώρα. Υπέρ. Υπέρ κατά. Απορρίφθηκε. Τέσσερα. Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και πάλι σε τμήματα ψηφοφορία, σε τρία τμήματα, έξι, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε, τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε, η εφτά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε, η εννέα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε, η δέκα υπέρ, κατά, Αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε στην Γιούρι τώρα, νομική επιτροπή. Δύο Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Η τρία Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ναι, θα ελέγξουμε λοιπόν την τρία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Γιούρι. τρία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. 29 υπέρ. Ένας εναντίον βλέπετε μάλιστα φίλοι μου. Λοιπόν, υπεψηφίστηκε. Πάει ναι, παραπονούνται ότι πάω πολύ γρήγορα, δεν γίνεται διαφορετικά, είναι βαρετή η δουλειά. Τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πέντε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Έξι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Εφτά υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. εννέα υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 12 υπέρ 12. 12 υπέρ. 12 συνεχίζουμε κύριοι. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Λοιπόν, τώρα μπορούμε 14, 15, β, γ, δ να τα πάρουμε όλα από κοινού. Λοιπόν, όσοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ε υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε F υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε G υπέρ γε κατά αποχές εγκρίθηκε λοιπόν τέλος ψηφοφορίας τώρα Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τελική ψηφοφορία όσοι είναι υπέρ τη έκθεση, παρακαλώ. Τελική ψηφοφορία. Α, εδώ βρίσκεται, Μαρία. Μαρία, er εδώ κάθεται αυτό. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Αποτέλεσμα 26 υπέρ. Δύο αποχές. Καμία ψήφος εναντίον. Ευχαριστούμε την Μαρία Σάντσες και τους Σκιώδη. Ευχαριστούμε. Έχω μια ερώτηση. Λοιπόν, έχουμε ακόμα δύο ψηφοφορίε, αλλά έχουμε τον κύριο Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ εδώ. Θέλετε να συνεχίσουμε τι ψηφοφορίε και μετά να εξαφανιστείτε και να μην ακούσετε τι θα πει ο κύριο Μαρτίνεθ. <laughs> Να συνεχίσουμε, τι λέτε. Αλλά παρακαλώ μετά να παραμείνετε στην αίθουσα, έτσι. Να μην φύγετε. Δεν θα ήταν ευγενικό αν εγκαταλείπαμε τον κύριο Μαρτίνεθ μετά τι ψηφοφορίε. Κυρία Μπεζιά, παρακαλώ, έχετε τον λόγο που Αποσύρω την τροπολογία μου αριθμός 16, παρακαλώ. Yes, yes, Thank you, Chair. Um, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία ήταν η έκθεση αυτή που ετοίμασα. Πιστεύω ότι είναι μια χρήσιμη έκθεση Ξέρουμε ότι έχει και τις προτεραιότητες της η Προεδρία. Να ξέρετε πάντως ότι ήταν πολύ επιτυχής η συνεργασία μας και ευχαριστώ και τους σκιώδεις εισηγητές και το προσωπικό και όλους τους ειδικούς επιστήμονες, υπερογνώμονες με τους οποίους συνεργαστήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Πολύ καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. 22 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Προφορική τροποποίηση 1 υπέρ κατά Αποχές εγκρίθηκε. 31. 31, όχι. Πάει αυτή. Συμβασμός 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 33, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 35, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 34, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 38, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Προφορική τροποποίηση 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 40 υπέρ υπέρ <laughs> υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 40 άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας τώρα αποτέλεσμα 17 υπέρ 10 εναντίον εγκρίθηκε 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 42 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 47 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τι είναι εδώ η τροπολογία 3 υπέρ, προφορική τροποποίηση 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Προφορική τροποποίηση 4 τώρα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 56 λοιπόν τώρα και 57 ταυτόσημες υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκαν. 58 υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε την 58, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 15 υπέρ 12 εναντίον εγκρίθηκε. 59 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 68, 69 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκαν 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 72 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε ναι να ελέγξουμε ωραία λοιπόν ψηφίζουμε άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 72 τέλος ψηφοφορίας αποτέλεσμα απορρίφθηκε 17 εναντίον 10 υπέρ απορρίφθηκε όπως είχα πει 73 υπέρ υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε που πάμε τώρα 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 78-79 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές. Άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 78-79. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 12 υπέρ 13 εναντίον απορρίφθηκαν. Πάμε στην 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 82-83 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκαν. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 89 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 90 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 90 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 14 υπέρ 12 εναντίον εγκρίθηκε τροπολογία 3 3 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε προφορική τροποποίηση 5 υπέρ τι λέτε συγγνώμη ε, λάθος ωραία η 4 πρώτα η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 5 τώρα προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 6 τώρα υπέρ κατά Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 6 ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα ισοψηφία 13-13. Απορρίφθηκε. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 9 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 11 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 15 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 16 υπέρ αποσύρθηκε η 16. Η 15, 15, 15 υπέρ Μα την ψηφίσαμε πριν, έτσι. Και η 16 αποσύρθηκε. Αυτό εννοούσα, μάλιστα. Έχει αποσυρθεί η 16. Και τώρα πάμε στη 17. 17 λοιπόν, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 19 και 20 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. Και 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν την 21 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα 12 υπέρ 15 εναντίον απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. Τι έχουμε τώρα, τροπολογία 1, εισηγητού, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Η 2, υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα 27 υπέρ. Καμία ψήφος εναντίον, καμία αποχή. Μάλιστα. Εσείς κύριε Σβέρ, θέλετε να πείτε κάτι. Κύριε Σβέρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου τη κυρία Χάνεμπολ, θέλω να... Μάλλον, ω και όντως θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Χάνεμπολ για την καλή συνεργασία που είχαμε μαζί. Έτσι καταφέραμε να πετύχουμε μια ωραία συμφωνία. Δείχνει αυτό ότι διαφορετικέ πολιτικέ ομάδε μπορούν κάλλιστα πολύ καλά να συνεργαστούν μαζί του. Υπέροχα. Εδώ ο κόσμο είναι ακόμα, θα έλεγε κανεί, ολόκληρο. Και περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία. Σαμπίνε, τι γίνεται. Πολύ σύντομη θα είναι η ψηφοφορία αυτή κύριε Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ. Εντάξει. Λοιπόν. Η κυρία Μπεναράμπατου. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας. Τους ευχαριστώ. Ωραία, ξεκινάμε. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε συμβιβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 6 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 8 καταπίπτει 6 δεύτερο τμήμα σε τμήματα. Πού είναι το σε τμήματα ψυχή. Είναι το δεύτερο τμήμα σε τμή, ως τμήμα. Ωραία. Καταπίπτει όμως τώρα, όχι. Α, η οκτώ καταπίπτει. Εντάξει. Τροπολογία 6 λοιπόν, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Μάλιστα. Καταψηφίστηκε, απορρίφθηκε. Η εννέα Υπέρ. Η δέκα καταπίπτει, έτσι. εννέα τώρα λοιπόν. Α, είχε απορριφθεί. Α, εντάξει, σίγουρα. Πολύ καλά. Λοιπόν, η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 9 υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 9. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 14 υπέρ 11 εναντίον. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ταυτόσημες. Η ε, 15 και 16 υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Υπήρχε κάποια διαφορά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε 15 και 16. Τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 18 υπέρ, 7 εναντίον εγκρίθηκαν αυτές. 14 υπέρ. Συμβιβασμός 2 λέτε. Α, εντάξει, συνεχίζουμε, περνάμε στο συμβιβασμό 2. Εντάξει, συμβιβασμός 2 λοιπόν, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ωραία, πού πάμε τώρα, 21. 21 σε τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα της 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 22, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα Απορρίφθηκε. 13 εναντίον, 11 υπέρ. Απορρίφθηκε. 23 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Ψηφίζουμε την 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 14 εναντίον 12 υπέρ απορρίφθηκε. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχέσα εγκρίθηκε 33 υπέρ κατά αποχέσα εγκρίθηκε και τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 26 υπέρ καμία ψήφος εναντίον καμία αποχή συγχαρητήρια θερμά κυρία Μπαναραμπατού Can I ask you please to stay a little bit because we have... Παραμείνετε παρακαλώ στις θέσεις σας γιατί έχουμε τον Αντιπρόεδρο Μαρτίνες Μαρτίνες τώρα, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την κατάσταση όσον αφορά τον ε, οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας. It's very interesting. Everybody can stay because uh, they can learn something. So,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 πιέζει υπέρ του σχεδίου αυτού. Υπάρχει και απόφαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ξέρουμε ότι προχωράει το σχέδιο. Ο κύριος Μαρτίνες όμως θα μας εξηγήσει πιο συγκεκριμένα πού βρισκόμαστε. Γιατί αν δεν ενδιαφερθούμε εμείς για αυτό το σχέδιο, ποιος θα ενδιαφερθεί. Γι' αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω πολλοί αριθμούς. Ελπίζω να μην αποχωρήσετε πριν ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Μαρτίνες. Ο κύριος Μαρτίνες Μαρτίνες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ειλικρινά ήταν πολύ ευχαριστώ για μένα που παραβρέθηκα στην ψηφοφορία και είδα πώς λειτουργεί η Επιτροπή αυτή. Ζηλεύω, βλέπετε. Ζηλεύω όταν βλέπω πώς λειτουργείτε εσείς εδώ. Για να δούμε, ίσως σε μια τρίτη, τέταρτη ζωή, άμα ξανάρθουμε σε αυτή τη ζωή. Πάντως, ε, πολύ θα ήθελα να συνεργάζομαι με την Doris με ιδιαίτερη ικανοποίηση έρχομαι εδώ σήμερα στην Επιτροπή σας για να συζητήσουμε μαζί. Θέλω ευθύ εξ αρχής να ξεκαθαρίσω ότι είναι η τέταρτη φορά, τέταρτη φορά που έρχομαι εδώ στην Επιτροπή αυτή για να εξηγήσω και για να ενημερώσω του συναδέρφους, τις συναδέρφους της Επιτροπής αυτής για το πώς προχωράμε. Και σας το λέω αυτό ευθύ εξ αρχής, διότι Τις στιγμές αυτές που ζούμε σήμερα, ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά που τίθεται είναι μήπως δεν υπήρξε αρκετή διαφάνεια, μήπως δεν υπήρξε αρκετή επικοινωνία, ενημέρωση. Θα επανέλθουμε σε αυτό και αργότερα. Πάντως, εδώ στην Επιτροπή αυτή έχουμε για τέταρτη φορά. Και μάλιστα μου το ζητάτε εσείς κάθε φορά και έρχομαι. Την προηγούμενη φορά Ήμουν εδώ τον Μάρτιο που μας πέρασε. Σημαντικά πράγματα είχαν συμβεί και τότε. Τώρα λοιπόν έρχομαι εδώ, πρώτον για να σας ενημερώσω, δεύτερον για να μοιραστώ μαζί σας ε, τις ελπίδες μου, την ικανοποίησή μου, αλλά και κάποιες ανησυχίες που έχω. Και σε ένα βαθμό μάλιστα έρχομαι επίσης εδώ για να σας ζητήσω τη συμβουλή σας και για να ζητήσω τη στήριξή σας. Τη συμβουλή σας σημαίνει ότι θέλω το δικό σας προβληματισμό, το συλλογικό προβληματισμό, μετά από αυτά που θα σας εξηγήσω και στη συνέχεια θέλω την βοήθειά σας, γιατί χρειαζόμαστε βοήθεια αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, εδώ που βρίσκεται το σχέδιο. Δεν θα χασομερίσουμε πολύ με το, τα προηγούμενα, πώς ξεκίνησε το σχέδιο κτλ. Υποθέτω ότι το γνωρίζετε πολύ καλά. Ξέρετε επίσης πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται για μια μακρά διαδικασία. Δύο στοιχεία θα σας ε, μεταφέρω μόνο για το τι έχει προηγηθεί. Πρώτον, υπάρχει μια έμπνευση, ένα σημείο από το οποίο ξεκινάει η έμπνευση για κάθε, για σχέδιο. Και εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας εμπνέεται από τον αντίστοιχο γερμανικό οίκο Ιστορίας που βρίσκεται στη Βόνη. Εγώ πρόεδρο, όταν ήμουν πρόεδρο μάλλον της ε, συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπη, ε, έδινα το βραβείο για τα μουσεία της Ευρώπης. Και με ιδιαίτερη συγκίνηση και ελπίδα επισκεφθήκαμε τα διάφορα μουσεία και πήγαμε μετά και στη Λιψία και καταλήξαμε να εμπνευτούμε από αυτό και να πούμε ότι θα έπρεπε να επαναληφθεί αυτό το εξαίρετο πείραμα, αυτή η εξαίρετη προσπάθεια και σε άλλες χώρες και σε άλλα επίπεδα. Δεύτερον, υπήρχε συνείδηση από την αρχή ότι ήταν αναγκαίο να διδάξουμε στις νέες γενιές, αλλά και σε λιγότερο νέες, σε Ευρωπαίους και σε μη Ευρωπαίους, να διδάξουμε λοιπόν αυτό που εγώ ορίζω ως το θαύμα που είναι μία Ήπειρος η οποία έζησε 20 αιώνες με κατοχές, με αδιαλαξίες, με ολοκληρωτισμούς, χρησιμοποιώντας τη βία και τον πόλεμο για να λύσει διάφορες διαφορές που υπήρχαν μεταξύ γειτόνων. Ε, λοιπόν, αυτή η Ήπειρος μέσα σε λίγες δεκαετίες μεταμορφώθηκε και έγινε ένα σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο για την συνύπαρξη, για την ολοκλήρωση, για την ε, ανοχή, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το διάλογο και για τη διατησία προκειμένου να λύνονται οι ίδιες διαφορές, οι οποίες πριν από λίγο καιρό τις λύναμε με τη βία. Αυτό είναι ένα θαύμα. Είναι θαύμα να μπορέσουμε να περάσουμε από την αντιπαράθεση στην ολοκλήρωση. Από τον ολοκληρωτισμό στη δημοκρατία. Και από τον πόλεμο στην ειρήνη. Είναι ένα θαύμα το οποίο μάλιστα δεν μας έρχεται από τον Θεό, είναι το θαύμα της πολιτικής και των πολιτικών στην υπηρεσία των λαών. Τη στιγμή λοιπόν που οι πολιτικοί δεν χαίρουμε ιδιαίτερης ε, εκτίμησης μερικές φορές. Ε, λοιπόν, καλό θα ήταν να διδαχτούν οι νέες γενιές, η κοινή γνώμη, και να μάθει ότι το θαύμα αυτό έγινε πραγματικότητα. Να μάθουν ότι πρόκειται επίσης για ένα θαύμα το οποίο δεν έχει παγιωθεί μια για πάντα. Είναι ένα θαύμα που χρειάζεται προσπάθεια για να διατηρηθεί, για να μην πάει πίσω, να μην σβηστεί. Γιατί από τη στιγμή που γίνεται πραγματικότητα, που έγινε μάλλον πραγματικότητα μέχρι τη σημερινή στιγμή, υπήρξαν ε, κομμάτια της ε, Υπήρου αυτής που για δεκαετίες δεν είχαν την ευκαιρία να χαίρουν των ίδιων ελευθερίας που έχερε ένα άλλο τμήμα της Ευρώπης. Μιλάω βέβαια για την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Υπήρχαν ε, άνθρωποι που ζούσαν στο ελεύθερο κομμάτι και άλλοι που ζούσαν κάτω από ανυπόφορες δικτατορίες. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος και η έμπνευσή μας για τον οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Τώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέθηκαν φυσικά πολλά ερωτήματα, πολύ λογικά. Το πρώτο ήταν γιατί, για ποιο λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία. Βρίσκω λογική την απορία αυτή. Βλέπετε τα κοινοβούλια δεν φτιάχνουν μουσεία συνήθως. Η απάντηση είναι εξή. Ξεκινάει το κοινοβούλιο και μπαίνει στην διαδικασία αυτή μετά από πρωτοβουλία του Χανς Πέτερ γιατί μάλιστα 15 χρόνια κράτησε η διαδικασία μέχρι να αποφασιστεί η δημιουργία. Ε, συστηματικά αποτύχαινε αυτή η ιδέα. Και αποτύχαινε γιατί είχαμε πολλούς μάγειρες μέσα στην ίδια κουζίνα. Στην αρχή του σχεδίου υπήρχε το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, η Βελγική Κυβέρνηση, το Άγιο Πνεύμα και δεν συμμαζεύεται. Ε, κάποια στιγμή λοιπόν έπρεπε να αλλάξουν τα πράγματα γιατί κάθε φορά όταν φτάναμε στο διατάφτα σταματάγαμε. Έπρεπε να υπάρξει συμφωνία Καμία χώρα δεν συμφωνούσε για το πού θα ήταν, η κάθε χώρα ήθελε τη δικιά της ιστορία. Ναι, αλλά εμείς δεν θέλαμε αυτό, δεν ήταν αυτό το σχέδιο, το αντίθετο ήταν. Αφού λοιπόν ε, αποτύχαμε πολλές φορές, κάποια στιγμή κάποιοι αρωματιστές αποφάσισαν ότι μόνο το Κοινοβούλιο εξαιτία της ίδιας του της φύσης μπορεί να προωθήσει ένα τέτοιο σχέδιο και να αντιμετωπίσει ό,τι δυσκολίες προκύψουν γιατί είναι μεγάλο στόχος για το Κοινοβούλιο. Εμείς ε, εκφράζουμε έναν πλουραλισμό εδώ. Μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προκλήσεις. Ε, μπορεί. Και αυτό αποδεικνύεται τώρα. Δεν θέλω να μπω από την άλλη μεριά στις άλλες λεπτομέρειες, γιατί εμείς και όχι Κομισιόν, για παράδειγμα. Ε, γιατί το Κοινοβούλιο μπορεί να αποτελέσει εγγύηση για την επιτυχία αυτού του σχεδίου. Μόνο το Κοινοβούλιο έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Εντάξει, η Επιτροπή από τη στιγμή ασχολήθηκε, η βελγική κυβέρνηση των Βρυξελών κτλ. Ο καθένας από αυτούς προσπάθησε να φροντίσει να παρέμβει. Η ευθύνη η βασική όμως ήταν η ευθύνη χρηματοδότησης από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό βέβαια δημιουργεί άλλα ερωτήματα. Γιατί, μήπως υπήρχαν άλλες αναλλακτικέ. Πάντως από την προηγούμενη φορά που βρέθηκα εδώ, μπορώ να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Και για αυτή την πρόοδο θέλω να σας ενημερώσω, που είναι και πηγή ικανοποίησης για μένα. Ένα από τα πράγματα στο οποία προχωρήσαμε ήταν το εξή. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν δύο διαδικασίες οι οποίες παράλληλα προχωρούσαν. Η μία διαδικασία είχε να κάνει με την επιλογή της επιστημονικής ομάδας η οποία θα αναλάβει να δημιουργήσει το μουσείο αυτό καθ' αυτό. Εννοείται πάντα υπό τον έλεγχο και την παρακολούθηση της Επιστημονικής Επιτροπής κλπ. Πάντως στην επιλογή του προσωπικού πρέπει να σας πω ότι ακολουθήσαμε μία μακρά διαδικασία και μία περίπλοκη διαδικασία. Πρέπει να σας το πω, αν και σας το λέω off the record αυτό, ότι η διαδικασία αυτή πέρα από το ότι ήταν μακρά και περίπλοκη από τη φύση της, ήταν ακόμα πιο περίπλοκη γιατί εδώ υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Μερικές φορές τρομερή και υπερβολικά δύσκολο να την ξεπεράσουμε γιατί συμμετέχουν και οι υπάλληλοι. Όταν νομίζεις ότι έχει ελέγξει το μηχανισμό, αν δεν, πρέπει πάντα να έρθει κάποιος ο οποίος σου ζητάει μια άδεια, κάποιος άλλος που πρέπει να υπογράψει και όταν έχει υπογράψει δεν έχει υπογράψει ο τρίτος και το καθεξής. Φτάνεις δηλαδή σε μια στιγμή που τρελαίνεσαι. Γιατί δεν βλέπεις την έξοδο από το τούνελ. Είναι η, ο λαβύρινθος της γραφειοκρατίας. Εν παρά τον λαβύρινθο αυτό όμω καταφέραμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη διαδικασία επιλογής με εκατοντάδες εκατοντάδες υποψηφίους τόσο για τη θέση του διευθυντή, της διευθύντριας ουσιαστικά του μουσείου, όσο και της επιστημονικής ε, ομάδας. Πράγματι ήταν περίπλοκη η διαδικασία, γιατί είχαμε πολλούς υποψηφίους. Και πρέπει επιπλέον να σας πω ότι το ότι είχαμε πολλούς υποψηφίους για τις νέες, νέα δέκα θέσεις επιστημόνων που θα βοηθήσουν. Εκεί είχαμε ιδιαίτερα ψηλή ποιότητα, για την διεύθυνση ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί, γιατί θέλαμε κάποιον που να έχει εμπειρία στα μουσεία, να είναι αναγνωρισμένος ιστορικός. Η ιστορική, έτσι, μιλάμε για άντρα γυναίκα. Και επιπλέον θέλαμε και κάποιον που να γνωρίζει και ξένες γλώσσες να έχει κάποια συγκεκριμένη ηλικία, γιατί είχαμε κάποιους εξαίρετους υποψηφίους, αλλά η ηλικία τους δεν τους επέτρεπε. Έχεις τρία χρόνια να φτιάξεις το μουσείο, άλλα τρία χρόνια για να αρχίσει να λειτουργεί, και μετά θα πάρει σύνταξη. Ε, όχι. Γι' αυτό, επειδή υπήρχαν δηλαδή πολλές προϋποθέσεις, πολλά κριτήρια, δυσκολευτήκαμε, αλλά καταφέραμε να κάνουμε μια εξαίρετη επιλογή που είναι εκείνη της κυρίας Φοφ ε, Γκάλ. Και μάλιστα θα σας πρότεινα να την καλέσετε εδώ κάποια μέρα. Να έρθει και να μιλήσετε μαζί της. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία του σχεδίου μας. Αν, έρθετε, αν την καλέσετε λοιπόν θα μπορέσετε να συζητήσετε μαζί της για το περιεχόμενο. Εμείς δεν ασχολούμαστε τόσο με το περιεχόμενο, αυτό είναι δικιά της ευθύνη. Πιστεύω θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι από τη Σλοβενία, αλλά έχει και κάποιες ολλανδικές ε, ρίζες. Ήταν και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην ε, διεύθυνση της Επιτροπής που αποφασίζει για το Ευρωπαϊκό Βραβείο για τα Μουσεία. Ε, ήταν στο Μουσείο της Λουμπλιάνας, ε, το οποίο έχουμε επισκεφθεί όλοι και έχουμε θαυμάσει. Αυτή λοιπόν είναι επικεφαλής. Είχαμε τώρα και μια δεύτερη επιτυχία. Σας έχουν μοιραστεί νομίζω κάποια, κάποιες φωτογραφίες. Πρόκειται για την επιλογή του αρχιτεκτονικού σχεδίου ξεκινήσαμε από την ιδέα ότι έχουμε το κτίριο Eastman, που είναι ένα κτίριο εδώ στο πάρκο, στο ίδιο πάρκο, στο οποίο είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παλιά ήταν ε, σχολείο δοντιατρικής που είχε φτιάξει κάποιος φιλάνθρωπος για φτωχά παιδιά στις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα. Έχω ακούσει τους διάφορους αρχιτέκτονους. Πολλοί λέγανε ότι δεν ήταν καλό. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλό γιατί βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, είναι όπως είναι και έχει και το πλεονέκτημα να είναι κάπως ιδιαίτερο χωρίς όμως να θεωρείται πολιτιστική, ιστορική κληρονομιά και να μην μπορεί κανείς να το αλλάξει. Δηλαδή επιδέχεται ορισμένες παρεμβάσεις το κτίριο αυτό καθ' αυτό. Επικοινωνήσαμε με όλες τις σχολές αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη και εκτός, κάπου 130 ε, ζήτησαν πληροφορίες. Από τους 130, 26 εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Από τους 26, 12 επιλέχθησαν ως φερέγγι εξαιτία της εμπειρίας του των σχεδίων που έχουν ήδη πραγματοποιήσει κτλ. Οι 12 αυτοί λοιπόν υπέβαλαν ένα προπροσχέδιο με κάποια σχέδια δικά τους. Υπέβαλαν λοιπόν κάποια σχέδια και από αυτά τα προπροσχέδια που υπέβαλαν μεγάλοι αρχιτέκτονες Ευρωπαίοι και μη Ευρωπαίοι, συζητήσαμε επί μακρό και αποφασίσαμε ότι έξι από αυτούς είχαν τα καλύτερα σχέδια και από αυτούς τους έξι καταλήξαμε σε δύο. Ορισμένοι πιστεύουμε ότι ο ένας έπρεπε να επιλεχθεί, άλλοι επαγγελματίες είπαν ότι έπρεπε να επιλέξουμε δύο. Και αυτό γιατί μετά θα γινόντουσαν διαπραγματεύσεις. Θα έπρεπε να καλέσουμε δηλαδή τους δύο καλύτερους για να συζητήσουμε μαζί τους. Αν ήταν μόνο ένας, ε, θα ήταν δύσκολο να μας προτείνουν όσο γίνεται καλύτερες τροποποίησεις, ενώ αν είναι δύο και είναι σε ανταγωνισμό μεταξύ τους, θα φροντίσουν να μας παρουσιάσουν τις καλύτερες δυνατόν τροποποίησεις για να τους διαλέξουμε. Και έτσι έγινε. Είπαμε, αν είχαμε καταλήξει σε έναν... Α, εσείς έχετε μόνο του ενός τις προτάσεις. Εντάξει, γιατί ένας επιλέχθηκε τελικά. Πάντως, όταν μας ήρθαν οι δύο επικρατέστεροι, εντυπωσιαστήκαμε από το επίπεδο, την ποιότητα. Ένας βέβαια τελικά κέρδισε. Είναι μια εταιρεία που κυρίως δρά στο Παρίσι, αλλά όχι μόνο και αλλού. Έκανε ας πούμε η εταιρεία αυτή το μουσείο του Πετυπαλέ στο Παρίσι, στην Τουλούζη. Μεγάλο κύρος έχει η αρχιτεκτονική, αυτό το αρχιτεκτονικό γραφείο. Άρα λοιπόν δύο μεγάλες επιτυχίες για τις οποίες εκφράζω την ικανοποίησή μου και που με γεμίζουν ελπίδα. Όμως χρόνος... ανέλπιστα, βρισκόμαστε μπροστά και σε κάποια εμπόδια, τα οποία είναι λογικό να τα έχουμε μπροστά μας. Άλλοι δεν το θεωρούν τόσο λογικό. Όπως και να έχει το πράγμα, τα προβλήματα πρέπει να τα εξετάζουμε σε βάθος και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις ικανοποιητικές για όλους λύσεις. Τα εμπόδια που έχουμε μπροστά μας έχουν να κάνουν καταρχήν με το οικονομικό ζήτημα και με κάποια θέματα αρχών επίσης. Ας ξεκινήσουμε από το δημοσιονομικό. Η κυρία Τρούπελ θα μας τα πει μετά, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην υπόθεση αυτή. Ποια είναι αυτά τα οικονομικά ζητήματα. Είναι ότι πέρυσι στον προπολογισμό του 2010 είχαμε ήδη συμπεριλάβει εκατομμύριο ευρώ κάτι τέτοιο. Το 2011 όμως υπάρχει ένα τμήμα 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που είναι μέρος του κόστους του σχεδίου που θα φέρουν σε πέρας οι αρχιτέκτονες. Επειδή μας είπανε μέχρι 3 εκατομμύρια θα χρειαστούν. Αυτό το τμήμα εγκρίνεται με τον προπολογισμό του 2011, αλλά μετά από παρεμβάσεις διαφόρων συναδέρφων και με στήριξη και της κυρίας ε, Τρούπερ, που ήταν η συγγήτρια για τον προπολογισμό, το ποσό αυτό μπαίνει στο αποθεματικό. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή Προπολογισμών έχει ε, κάποιες, ε, κάποια ερωτήματα, ένα, δύο, τρία, και μόνο όταν πάρει απαντήσεις και διευκρινήσεις στις απορίες της αυτές θα μπορέσει να εκταμιευτεί το ποσό αυτό. Λογικό. Είναι στο ποθωματικό προς το παρόν. Δεν είναι όμως αυτό το μόνο εμπόδιο <clears throat> και παρά τόσα πιστεύουν πολλοί συνάδελφοι που συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό, εγώ καταλαβαίνω τα προβλήματα της Επιτροπής Προϋπολογισμών που δεν είναι μόνο πού θα πάνε τα χρήματα αυτά. Υπάρχουν δύο ακόμα κεφάλαια απορριών που θεωρώ επίσης αιτιολογημένα. Το πρώτο είναι πόσο τελικά θα στοιχήσει αυτό το σχέδιο. Μέχρι να ανοίξει δηλαδή το μουσείο. Πόσο θα μας κοστίσει. Λογική απορία. πρέπει να έρθει ή όχι το αποθεματικό των 2,5 εκατομμυρίων. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία απορριών. Πόσο θα στοιχήσει η λειτουργία του μουσείου στη συνέχεια. Αφού ξεκινήσει το 2014, όταν θα έχει κλείσει ένα αιώνα από την ε, λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρώτον λοιπόν πώς θα χρησιμοποιηθούν τα 2,5 εκατομμύρια. Δεύτερον πόσο θα στοιχήσει συγκεκριμένα και αιτιολογημένα και με επιχειρήματα το όλο σχέδιο μέχρι να ανοίξει το μουσείο. Και τρίτον πόσο θα στοιχήσει η λειτουργία του μουσείου αυτού. Κατά τη γνώμη μας έχουν δοθεί όλες οι πληροφορίες και πρέπει και να σας ομολογήσω με κάποια θλίψη ότι πολλές φορές αντιμετωπίσαμε συναδέρφους οι οποίοι έρχονται και ζητάνε πληροφορίες για στοιχεία τα οποία τους έχουμε ήδη δώσει. Τα έχουνε, δεν διάβασαν τα χαρτιά. Ή δεν ήταν παρόντες όταν τις δώσαμε αυτές τις απαντήσεις. Ε, αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί κάποιον εκνευρισμό. Τρεις φορές που πήγαμε, ο κύριος Πέτερινγκ και εγώ, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Στη διάσκεψη των Προέδρων Πολιτικών Ομάδων. Και στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιουργήθηκε δυσλειτουργία. Διότι στη διάσκεψη Προέδρων Πολιτικών Ομάδων υπήρξε ενθουσιασμός και από όλη τη στήριξη του σχεδίου και των δεδομένων και του προπολογισμού που ζητήσαμε, που προβλέπετε. Ενώ στην Επιτροπή Περιπολογισμών υπήρξε μια ένταση και υπήρξε μια παράδοξη κατάσταση. Ορισμένοι συνάδελφοι λένε «Α, εμεί δεν ξέρουμε τίποτα από όλε αυτέ τι πληροφορίε, δεν έχουμε κανένα στοιχείο» και σηκώνεται άλλο συνάδελφο τη ίδια, κοινοβουλευτική επιτροπή, για να απαντήσει με όλα τα στοιχεία που ο προηγούμενος δεν είχε. Και σηκώνεται κι άλλο με τα χαρτιά και λέει «Να, την πληροφορία αυτή την έχετε στου φακέλου σα. Διαβάστε το. Αν το είχατε διαβάσει, θα ήσασταν ενημερωμένοι. Βλέπετε, αυτή είναι η πραγματικότητα του πώς λειτουργούμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι η έκθεση που σας δίνω, εντάξει, δεν είναι μόνο κάτι που μου έχει ετοιμάσει η γραμματεία, είναι τα στοιχεία που έχουμε. Αν λοιπόν ακούγονται κατηγορίες ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, η απάντηση είναι ότι από την αρχή μέχρι το τέλος η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και οι άλλοι τα έχουν τα στοιχεία. Αλλά δεν φτάνει γιατί έρχεται και ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών ο οποίος δεν ενημερώθηκε ατομικά, ενημερώθηκε ως πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Και η κυρία Πάκ όταν ήρθε στις συναντήσεις αυτές για να ενημερωθεί ήρθε ως πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και αναλαμβάνει την ευθύνη να σας ενημερώσει. Και η κυρία Πακ μας ζήτησε τέσσερις φορές να έρθουμε εδώ. οι επιτροπές δεν μας το ζήτησαν καθόλου. Έτσι λοιπόν, σήμερα ευτυχώς έχει απελευθερωθεί το ποσό που ήταν στο ποθηματικό των 2,5 εκατομμυρίων και έτσι ξεκινήσαμε με τα συμβόλαια με τους αρχιτέκτονες και ξεκινάμε και βελτιώνεται η κατάσταση. Αλλά υπάρχουν και άλλα να γίνουν για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Δεν είναι μόνο το θέμα των ε, ποσών, να ξέρουμε ακριβώς πόσο θα στοιχήσει η ολοκλήρωση του μουσείου, η λειτουργία του μουσείου κλπ. Και σας θυμίζω ότι σε κάποια από τις συνεδριάσεις που έχουμε πάει, ορισμένοι συνάδελφοι, χωρίς να έχουν κανένα σημείο αναφοράς, σηκώνονται και σου λένε από την εμπειρία μου εγώ ξέρω ότι όταν λέτε ότι θα στοιχήσει 50 εκατομμύρια θα στοιχήσει 100. Το έχουμε ακούσει αυτό. Είναι τοποθετήσεις που είναι αέρας κομπανιστός. Δεν ξέρω αν στις χώρες τους έτσι γίνονται τα πράγματα. Ε, σε χώρες δεν γίνονται, πρέπει να τους πούμε. Και όταν δίνουμε κάποια στοιχεία, αυτά τηρούνται. Μέρη Τερέσα, ξέρει πολύ καλά για τι πράγμα μιλάω, έτσι. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια, ώστε τα ποσά τα οποία προτείνουμε για το άνοιγμα του μουσείου είναι πολύ λογικά και πολύ συγκεκριμένα, έχουν βάση. Ίσως είναι πιο δύσκολο να δώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πόσο θα στοιχήσει η λειτουργία του μουσείου στη συνέχεια. Αλλά υπάρχουν κατέτος ποσά. δεν είναι γελία. Αν τα συγκρίνουμε με το πόσο στοιχίζει η λειτουργία ενός μουσείου στις χώρες μας. Για να ανοίξει το μουσείο, λέμε ότι θέλουμε 12-13 εκατομμύρια στον προπολογισμό του 2012, 20-22 για το 2013 και 14 15 για το 14. Διότι πρέπει να ενισχυθεί ο σκελετός του κτηρίου, να γίνουν δηλαδή διάφορα ε, δομικά έργα, στατικά και πρέπει να υπάρχει ε, διάδραση με ένα σωρό οργανισμούς και όργανα από διάφορες χώρες και σε διάφορες γλώσσες που μας είπαν ότι θέλουν να συμμετάσχουν. Δεν πρόκειται μόνο για τη μόνιμη έκθεση, αλλά πρόκειται και για την άλλη η οποία θα μεταφέρεται, θα πηγαίνει στις διάφορες πρωτεύουσες ή για άλλες προσωρινές εκθέσεις που θα λαμβάνουν χώρα εκεί. Έτσι λοιπόν πώς ακριβώς θα στοιχήσει η λειτουργία, είπαμε περίπου 13 εκατομμύρια το χρόνο, αλλά αυτό είναι ένα ποσό που συζητιέται. Θα είναι ανοιχτό και το Σάββατο και την Κυριακή. Χρειάζεται λοιπόν ασφάλεια. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα έξοδα πέρα από τα έξοδα που έχουμε συνήθως για τέτοιες περιπτώσεις. Και θα ολοκληρώσω με το εξή. Για μένα είναι σαφές ότι το σχέδιο αυτό δεν θέλει να γίνει μια γενική διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που θέλει είναι να γίνει κάτι το οποίο θα αυτοδιαχειρίζεται από ένα ίδρυμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει βέβαια λόγο. Ούτε θέλει το σχέδιο αυτό να βρίσκεται συστηματικά στον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η λειτουργία του δηλαδή. Μια από τις συζητήσεις που έγιναν και ήταν ιδιαίτερα έντονη ήταν γιατί δεν συζητάμε για χρηματοδότηση με την Κομισιόν και τις Βελγικές Αρχές. Ε, η απάντηση είναι δεν το κάνουμε γιατί τότε θα παρέλειε το σχέδιο. Πιστεύω όμως ότι όταν φτάσουμε στην λειτουργία, εκεί θα συμμετάσχει η Κομισιόν και θα συμμετάσχουν και οι βελγικές αρχές. Κάποιος είπε, ε, τώρα, όχι. Αν καταφέρουμε να ξεκινήσουμε ε, τη λειτουργία, θα βρούμε, θα βρούμε και σπόνσορες. Είτε ιδιώτες, είτε κάτι άλλο, οι οποίοι θα θελήσουν να συμμετάσχουν και να χρηματοδοτήσουν αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Και θα τελειώσω και με κάτι για το οποίο θέλω τις δικές σας ιδέες, τη γνώμη σας. Είναι αλήθεια ότι δεν ακολουθήσαμε τον καθαρά κοινοβουλευτικό δρόμο που θα ήθελα με μια έκθεση από μια κοινοβουλευτική επιτροπή επί της ουσίας και άλλες δύο όπου να γνωμοδοτούν και να συζητηθεί η έκθεση αυτή και εδώ και στην Ολομέλη κτλ. Δεν ακολουθήσαμε αυτό το δρόμο. Ομολογώ ότι μερικές φορές ε, το σκέφτηκα. Αλλά σκέφτηκα ότι μια τέτοια διαδικασία θα είχε οδηγήσει σε ένα σωρό προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερα αν συζητούσαμε με την Επιτροπή Πολιτισμού, με την Επιτροπή Προπολογισμών, να συμμετέχουν αυτές οι επιτροπές στο σχέδιο, αλλά να μην μπαίνουμε στη διαδικασία ψηφοφορίας. Εξάλλου στο Προεδρείο έχουμε ψηφίσει επανειλημμένα. Έχουμε ε, επίσης ψηφίσει επανειλημμένα στη διάσκεψη Προέδρων, όχι όμως στην Ολομέλεια. Γιατί εκεί θα κολλάγαμε. Στη συζήτηση πάντως που θα έχουμε θα συζητήσουμε για τον προπολογισμό του 2012. Και εκεί πρέπει να δούμε τι μηχανισμό θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου εκεί η Ολομέλεια να μπορέσει να αποφανθεί κάποια στιγμή. Έχω εμπιστοσύνη στους πρόεδρους των πολιτικών ναι. ομάδων. Αν οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων ομόφωνα λένε ότι στηρίζουν χωρίς επιφυλάξει το σχέδιο αυτό, ε, υποθέτω ότι όταν φτάσουμε στη ψηφοφορία οι πολιτικές ομάδες θα ψηφίσουν αντίστοιχα. Ωραία, σε ορισμένες ομάδες υπάρχουν επιφυλάξεις. Εγώ έρχομαι από μια ομάδα της αριστεράς, έτσι, της αριστεράς και έχουμε μια φιλοσοφία για την ιστορία πιστεύω ότι ως σημείο αναφορά η αριστερά περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον ε, έχει την ιστορία. Με αυτές τις ιδέες λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε και να συζητάμε με τους διάφορους. αν θα είναι πόσα, εντάξει θα το δούμε. Τώρα πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε και ζητάω τη γνώμη σας και τη στήριξή σας πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον μηχανισμό έτσι ώστε πραγματικά όσο γίνεται πιο γρήγορα να έχουμε την στήριξη της Ολομέλειας. Γιατί έτσι θα βγούμε από αυτή την αφησιμία στην οποία βρισκόμαστε και από ορισμένοι σηκώνονται και λένε δεν υπήρξε διαφάνεια, δεν συζητήθηκε, δεν έκανε, δεν έδειξε. Εσείς το ξέρετε ότι και συζητήθηκε και ψηφίστηκε και εγκρίθηκε το σχέδιο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Εδώ βρισκόμαστε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει. Αγαπητέ μου φίλε, με τέτοιες προσπάθειες που καταβάλεις δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει μαζί σου. Για ένα τέτοιο εγχείρημα με τόσους πολλούς αντιπάλους πρέπει να φλέγεται κανείς γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να υλοποιηθεί και για το βραβείο Λούξ όλα όσα έχουν σχέση με το όραμα και το όραμα της Ευρώπης το όραμα του Ρομπέρ Σιουμάν όλα αυτά σκεπάζονται και σβήνουν αν σκεφτόμαστε μόνο τη σημερινή, την καθημερινή δουλειά που πρέπει να την κάνουμε αλλά πρέπει να δουλεύουμε και για ένα όραμα ο οίκος της ιστορίας πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα πως το κοινοβούλιο μπορεί να συνεργαστεί να εργαστεί για ένα τέτοιο στόχο Συμφωνώ μαζί σου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τα χρήματα αυτά τα οποία δίνονται από εμά. Δεν χρειάζεται να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εγχείρημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι για τον πολιτισμό πολύ στενό. Έχουν διαφορετικέ απόψει για το τι πρέπει να καλυφθεί. Αν είναι μια ιδέα του Κοινοβουλίου, πρέπει το Κοινοβούλιο να μεριμνήσει από τα δικά του κονδύλια να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο. Βρισκόμαστε σε καλή πορεία. Πρέπει μόνο εδώ να διαφωνήσω σε ένα θέμα. Δεν το θέλω αυτό όταν είπες ότι ελπίζω ότι οι πρόεδροι των ομάδων, τι είπες, οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων είπες, Α, δεν με έχει κανένα, είπε στο χέρι. δεν μα έχει στο χέρι κανένα πρόεδρο κοινοβουλευτική ομάδα. Αγαπώ τον πρόεδρο τη ομάδα μου, αλλά κάνω αυτό το οποίο εγώ πιστεύω και είμαι όταν είναι οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων είναι υπέρ, λέει ο μιλητή. Ναι, αλλά δεν συμβαίνει αυτό πάντα, να είναι πάντα υπέρ. Γι' αυτό πρέπει να μεριμνήσουμε. Οι συνάδελφοι που δεν έχουν τέτοια μεγάλη σχέση με θέματα πολιτισμού θα είναι υπέρ αυτού του εγχειρήματο. Ήθελα να το αναφέρω αυτό. Και θα ήθελα λοιπόν εδώ σε σχέση με του συναδέλφου, ε, όσοι έχουν συνεργαστεί σε σχέση με, την ε, δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα μα εγκαταλείψει σε τον Απρίλιο διότι θα εργαστεί για τον οίκο τη ε, ιστορία, λοιπόν, τον Ευρωπαϊκό οίκο. Διότι θα είναι το αυτή μα, ε, το μάτι μα ε, στον οίκο τη ιστορία. Και έτσι μπορούμε να τη ευχηθούμε κάθε καλό και να ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε για το γεγονό ότι ήταν εδώ δύο χρόνια σε εμά, στη δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή, εργάστηκε εξαιρετικά, γέννησε και ένα παιδί εντωμεταξύ και θα περάσει στον οίκο τη ιστορία. Όλα τα καλά, αγαπητοί Κωνσταντσε. Και τώρα θα λάβει τον λόγο ο συνάδελφος Καβαντά. Κύριε Καβαντά, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Μιγγέλ για την παρουσίαση. Χαίρομαι που επιτέλους έχουμε κάποια στοιχεία πρόοδου. Θα μπω στην ουσία της υπόθεσης. Ακούσαμε πολλά τις τελευταίες εβδομάδες για τις κριτικές που έγιναν οικονομικές, η έλλειψη διαφάνειας, υποτιθέμενη έλλειψη διαφάνειας. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας, απειλείται από υπερβολική διαφάνεια. Να πω λοιπόν παρακαλώ δημόσια το εξής. Ζούμε σε μια εποχή δημοσιονομικής λιτότητας. Ναι. Παρόλα αυτά θα πρέπει να βρούμε κάποιες μορφές οικονομικής διαχείρισης αυστηρές έτσι ώστε να προχωρήσουμε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θεωρώ ότι είναι χρήσιμο. Δεύτερον, σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας μείνουμε στο πνεύμα των συνθήκων. Στόχος της Επιτροπής είναι η Γενική Γραμματεία των Οργάνων με πολιτικές αρμοδιότητες για τη διασφάλιση του κοινωνικού συμφέροντος, δηλαδή της λειτουργίας των οργάνων και των πολιτικών σήμερα και φυσικά μεσοπρόθεσμα. Θα θέλαμε άλλωστε και βράχει πρόθεσμα να ήταν κάπως πιο δραστήρια για το μέσο πρόθεσμο αυτοί που ασχολούνται με προβλέψεις και προοπτικές θα το φροντίσουν. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να επιβραδύνω ή να επιβαρύνουμε την λειτουργία του οργάνου μας με ένα άλλο όργανο το οποίο δεν είναι εκεί ο ρόλος του και νομίζω τα πράγματα είναι δύσκολα ήδη και δεν πρέπει να τα μπλέξουμε. Κάποια επιπλέον θετικά σημεία τώρα, τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, είμαι σίγουρος θα συμφωνήσετε μαζί μου. Είμαι ιδιαίτερα υπέρ του προγράμματος αυτού. Είμαι ιδιαίτερα υπέρ και της ομάδας που το προωθεί, όχι μόνο εσύ Μιγγέλ και οι φίλοι σου. Αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν μιλάω για τα πολιτικά θέματα, αλλά η προσωπική εμπλοκή και η εικόνα του Πέτερινγκ στη συγκεκριμένη ιστορία ε, νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενη και λόγω της δικής του ιστορίας, κάτι το οποίο απομακρύνει κάθε αμφιβολία για την ιστορική ειλικρίνεια ε, μοιράζομαι μια κοινότητα θα έλεγα μαζί του σε επίπεδο προοπτικής όταν ήμασταν μικροί αλλά η συμπεριφορά του όταν ε, μεγάλωσε, ενηλικιώθηκε, έγινε βουλευτής, πήρε ευθύνε, έγινε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα πνεύμα πολιτικής δεκτικότητας και ουδετερότητας όλα αυτά δείχνουν ε, και πρέπει να του δώσουμε την εμπιστοσύνη μας και ε, προσωπικά αυτό το κάνω. Σε 150 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ήπειρος ε, έκανε δώρο στον εαυτό της τρεις μεγάλους πολέμους, ολοκληρωτικά τυραννικά καθεστώτα, τρεις πολέμους εκ των οποίων οι δύο παγκόσμιοι. Αναφλέξαμε τον υπόλοιπο κόσμο δις και σαν να μην έφτανε αυτό, αυτοί οι πόλεμοι που προκάλεσαν εκατομμύρια νεκρών, που οδήγησαν όπως λέει η Χάνα Άρεντ στην αυτοκτονία την Ήπειρο αυτή, μετά από τους πολέμους ε, είχαμε τυραννικά καθεστώτα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ε, τυραννικά καθεστώτα, απολυταρχικά, ε, ναζιστικά, σταλινικά, ε, τυραννικά καθεστώτα στο Νότο, στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει αρκετά με αυτή την τρέλα, ας καταλάβουμε γιατί έγιναν όλα αυτά και όλα αυτά τα μηνύματα αταξίας τα οποία βιώνουμε σήμερα ας μην τα ξαναζήσουμε και τα σχολεία, η σχολική εκπαίδευση και τα παιδιά προς τα οποία προορίζεται η προσπάθεια αυτή να καταλάβουν τι έγινε. Στο Νότο τα τυραννικά καθεστώτα προκλήθηκαν από τους στρατιωτικούς. Στην Ανατολική Ευρώπη προηγήθηκε η κάλπη και μετά ακολούθησαν τα τεθωρακισμένα οι εκτοπισμοί και οι εκτελέσεις. Γι' αυτό είμαι υπέρ αυτού του προγράμματος, αυτού του σχεδίου, το μουσείο αυτό θα πρέπει στην ουσία να προσδώσει μια κοινή ταυτότητα στα παιδιά, τους νέους και τους έφηβους της Ευρώπης, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και αυτούς που έρχονται εκτός Ευρώπης. Ποια είναι αυτή η κοινή θρησκεία. Η ελευθερία, η δημοκρατία δεν θα καταστραφούν παρά μόνο αν δεν τις χρησιμοποιούμε και γι' αυτό ακριβώς το μουσείο αυτό θα πρέπει να μας οδηγεί στο σεβασμό των θεσμών και στην ε, συνεχή φροντίδα της δημοκρατίας. Τελειώνοντας. Ο Έλλη Βίζελ εδώ και λίγο καιρό όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου μας είπε ότι οι λαοί που δεν γνωρίζουν την ιστορία τους εκτίθενται στο να τη ζήσουν εκ νέου. Ε, μιλούσε σαν ιστορικός όταν το είπε. Όταν βλέπει κανείς την άνοδο των εξτρεμισμών στις δικές μας χώρες, οι οποίες ενθυμούνται φυσικά τι έχει συμβεί, νομίζω ότι ε, η φράση αυτή δεν είναι μία απλή ιστορική υπενθύμαση, στην ουσία είναι μία προφητεία και το Μουσείο της Ιστορίας πρέπει να μας πείσει να εξουδετερώσουμε αυτές τις συμπεριφορές. Αλλιώς θα σας θυμίσω τον Τσβάιχ, τεράστιος καλλιτέχνης, λογοτέχνης, δραματουργός, διηγηματογράφος. Ευρωπαίος πρώτα, Αυστριακός μάλλον πρώτα, Ευρωπαίος μετά, εβραϊκής καταγωγής, εξορίστηκε από τη Βιέννη στο Βερολίνο γιατί βρήκε την ελπίδα, έχασε την ελπίδα στο Βερολίνο, πήγε στην Αγγλία και έδωσε τον επικίδιο, εξεφώνησε τον επικίδιο λόγο του Φρόιντ και πήγε μετά στις Ηνωμένε Πολιτείε, κατέληξε στη Βραζιλία και στο τέλος του 42 αυτοκτόνησε κατανοώντας ότι η τρέλα των Ευρωπαίων καταστρέφει αυτή την Ήπειρο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα στηρίζω συστηματικά αυτό το προτινόμενο μουσείο και τα διαχειριστικά πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να θεωρήσω δεδομένο ότι όταν έχουμε μεγάλα προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν κάνουμε λόγο για θέματα κονδυλίων του προϋπολογισμού ή όταν έχουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο ε, μια και η πρόσθετη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα πολιτισμικά δεν είναι πάντα πιστικό επιχείρημα για τα κράτη-μέλη, μπορώ να πω τότε ότι οι πολίτες αν δεν γίνουν αυτά δεν θα μπορούν να δουν ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες και όλα αυτά πρέπει να αναφθούν στο ότι δεν τα καταφέραμε μέχρι σήμερα από κοινού να βρούμε και να δημιουργήσουμε αυτές τις κοινέ ευρωπαϊκές αξίες που θα ισχύουν πανευρωπαϊκά. Αν πάμε στη ΣΥΠΑ ή στην Ασία ή στην Αφρική τότε το βλέπουμε και το νιώθουμε ξεκάθαρα ότι έχουμε κοινέ ευρωπαϊκές αξίες εμείς ε, οι Ευρωπαίοι που μπορούν να πούν πολλά πράγματα στους άλλους και αυτό πρέπει να περάσουμε στις επόμενες γενναίες και αυτό να τους δώσουμε, να μεταλαμπαδεύσουμε. Αυτό το εγχείρημα θα ενισχύσει το εγχείρημα της οικοδόμησης της Ευρώπης σε ένα πολύ αποφασιστικό σταυροδρόμι, σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Τις κοινέ μας αξίες ε, ως Ευρωπαίοι πρέπει να τις έχουμε πάντα μπροστά μας, ως κληροδότημα της ιστορίας μας. Αν το κάναμε αυτό θα υπήρχαν λιγότερες αντιστάσεις. Οι κυβερνήσεις θα εργαζόντουσαν περισσότερο, θα συνεργαζόντουσαν περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ ενό κοινού εγχειρήματο. Και όταν πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια δεν θα υπήρχε αντίσταση, τόσο μεγάλη αντίσταση. Έχω υπόψη όχι μόνο τα θέματα τη Επιτροπή Πολιτισμού και μπορώ φυσικά να σα διασφαλίσω ότι θα υποστηρίξω το έτοιμά σα και στην Επιτροπή Πολιτισμού και στην Επιτροπή Προπολογισμών. Τώρα ίσως ένα ερώτημα ακόμα το οποίο πρέπει να δούμε αλλά σίγουρα υστερότερα θα ξανασυναντηθούμε στο μέλλον και θα ξανασυζητήσουμε τα θέματα. Αυτό το οποίο ζητήσατε ως συμβουλή και υποστήριξη η Επιτροπή Πολιτισμού θα εμπλακεί και θα υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα. Θα με ενδιαφέρε να ξέρω κατά πόσο μπορούμε να εργαστούμε, να συνεργαστούμε εμείς σε αυτό το εγχείρημα. Τι σημαίνει αυτό χειροπιαστά ότι θα θέλατε την συμβουλή μας και την υποστήριξή μας. Τι θα σήμαινε αυτό συγκεκριμένα χειροπιαστά χειροπιαστά. Επειδή με ενδιαφέρει άμεσα αυτό. Χάνιμπαλ παρακαλώ, κυρία Χάνιμπαλ. Είναι εξαιρετική ιδέα πιστεύω αυτή. Είναι κάτι το φανταστικό. Είναι ένα μεγαλόπνο όραμα να δημιουργηθεί αυτός ο οίκος ευρωπαϊκής ιστορίας και συμφωνώ με όλα όσα προαναφέρθηκαν. Και νομίζω ότι σίγουρα θα προχωρήσει, θα προαγάγει αυτά τα οποία εμείς στην Ευρώπη ζούμε και έχουμε ως ιστορία, ως αξίες. Υποστηρίζω απόλυτα αυτό το εγχείρημα. Είναι ωραίο να δει κανεί ότι εμπλέκεται πλήρως αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αν είναι κάποιου ή θα έλεγα κοντινό δικό του εγχείρημα είναι δικό μας όσο γίνεται πιο πολύ. Και τώρα κάποια πολύ χειροπιαστά θέματα θα ήθελα να αναφέρω Μιγγέλ. Ευχαριστώ βέβαια πάρα πολύ για τη δουλειά που έκανες. Έκανες εξαιρετική δουλειά για να επιτευχθεί αυτό και να προχωρήσει. Έκανες λόγο για να υπάρχει διάδραση, διαδραστικό πλαίσιο, να συμμετέχουν οι επισκέπτες και σε σχέση με τόσα πολλά θεσμικά όργανα και όλοι θα ενδιαφερόντουσαν να συμμετάσχουν, εμπλακούν και ότι είπες ότι για τα ίδια τα εκθέματα θα μπορούσαν να, ε, να, να μπορούν να ε, εκτίθενται ε, σε εκθέσεις ε, περιοδικά ανά την Ευρώπη. Θα με ενδιέφερε να ξέρω ποια θα ήταν αυτά τα εκθέματα. Κάνουμε και συζητάμε πολύ, κάνουμε λόγο για αυτό το όραμα, για αυτή την προσέγγιση την ιστορική. Το κτίριο είναι πολύ ωραίο. Με ενδιαφέρει πώς τα εκθέματα αυτά θα συντεθούν και πώς θα λειτουργήσουν αυτά. Τι θα βλέπουμε εμείς ε, σε αυτόν τον οίκο της ιστορίας χειροπιαστά. Και επίσης πώς θα ενθαρρυνθούν οι πολίτες, ή τα άτομα να πάνε και να επισκεφθούν αυτό τον οίκο της ιστορίας. Προφανώς έρχονται στις Βρυξέλλες οι επισκέπτες στο Ευρωκοινοβούλιο, επισκέπτονται το Ευρωκοινοβούλιο. Βρίσκεται εδώ, εντάξει. Όταν θα, είναι, θα γίνεται αυτό, για να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να προαχθεί, να το γνωρίσουν οι πολίτες και να το επισκέπτονται. Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα για αυτό το σκέλος, να μας ενημερώσεις παρακαλώ. Η κυρία Τρούπελ παρακαλώ. ναι σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα για το θέμα σύλληψης και προσέγγισης αυτού του οίκου της Ευρώπης να πω ότι εδώ και πολύ χρονικό ε, διάστημα ε, σε σχέση με αυτό το, τη μελέτη που έχουμε για το πώς θα ε, πάρει μορφή αυτός ο οίκος της ιστορίας, πώς η πολυμορφία της ευρωπαϊκής ιστορίας θα καλύπτεται γιατί δεν υπάρχει μία και μοναδική και μόνη ευρωπαϊκή ιστορία. Πώς η σύλληψη αυτή θα προχωρήσει είναι μια ιδέα που την υποστηρίζω απόλυτα. Έχει δίκιο η Ντόρις ότι βρίσκεται στη γραμμή του οράματος του Ρομπέρ Σιουμάν και των άλλων μεγάλων Ευρωπαίων. Εγώ ίδια συνέταξα μια έκθεση για τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στον οίκο του Ευρωπαϊκού, στο έτος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του 2009. Γι' αυτό γνωρίζω όλα τα επιχειρήματα υπέρ και γιατί είναι αναγκαίο οι επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα και δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα επιχειρήματα λοιπόν τα συμμερίζομαι όλα. Μια και είμαι συγγήτρια για τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2011 σε σχέση με τα προβλήματα του προϋπολογισμού που υπάρχουν, δεν πρέπει να τα υποτιμάμε αυτά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, με ένα ποσό 16 ε, ε, ε, εκατομμυρίων έχουμε μπροστά μας. Είναι περίπου ο προϋπολογισμός για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Δεν είναι αντεπιχείρημα κατά ενός νέου εγχειρήματος για τον οίκο ιστορίας. Θέλω όμως να πω ότι για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν θέλουμε μια τέτοια νέα προτεραιότητα, και το επαναλαμβάνω, υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά επειδή είναι περιορισμένη και τεταμένη η κατάσταση από πλευρά κονδυλίων, ο Λεβαντόφσκι απέστειλε μια επιστολή και είπε ότι το σύνολο του προπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου μόνο κατά 1% μπορεί να αυξηθεί. Αυτή τη στιγμή κάνουμε διαπραγματεύσεις ε, για τον προπολογισμό 2012 ως ομάδα και ως κοινοβούλιο ότι πρέπει το ποσοστό πληθωρισμού να λαμβάνεται υπόψη και να έχουμε και ε, την προσπάθεια σε σχέση με την αύξηση. Κάποιοι θέλουν να πάμε και στο 2%. Όμως κάποιοι έχουν καταλήξει στο 5,2% πάνω από αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουμε. Αν δημιουργήσουμε την εντύπωση στους πολίτες ότι την ανάγκη, τα δεινά, τον πόνο που ε, υφίστανται οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα αγνοούμε και θέλουμε να δαπανίσουμε μεγάλα κονδύλια για ένα τέτοιο εγχείρημα, δεν θα είναι αποδεκτό αυτό το εγχείρημα από τους πολίτες. Σήμερα το πρωί στη Stuttgart Zeitung, την εφημερίδα της Στουτγάρδης, υπήρχε ένα άρθρο όσον αφορά το νίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας για ένα αποθεματικό 2,5 εκατομμυρίων που απελευθερώνεται και τώρα θα πούν ότι παριστάνουν ότι έχουν όλα τα λεφτά του κόσμου δικά τους και δεν λαμβάνουν υπόψη καμιά ανάγκη λιτότητας. Και πρέπει να αντιδράσουμε πολιτικά σε τέτοιες θέσεις. Αν δεν έχουμε και δείξουμε πολιτική ευαισθησία, τότε πρόσθετα προβλήματα θα δημιουργήσουμε και θα καταλήξουμε να αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε και να πούμε αν είμαστε υπέρ αυτής της προτεραιότητας, όπως εγώ είμαι υπέρ, πρέπει κανείς να είναι πρόθυμος να εξοικονομήσει κονδύλια αλλού και να μην καταλήξουμε σε αυξήσεις που θα είναι υπερβολικές. Αυτό είναι πολιτικά η θέση μου. Και έχω το πρόβλημα με τους συναδέλφους μου λόγω αυτών το ότι μέχρι σήμερα δεν είναι πρόθυμοι να καταλήξουν σε εκταμιεύσεις και προτάσεις εξοικονόμησης ε, που θα οδηγούν σε κάποια οικονομία και περικοπές αλλού. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη αυτά αν είμαστε υπέρ μιας τέτοιας νέας προτεραιότητας όπως τον οίκο της Ευρώπης και να είμαστε πρόθυμοι να σκεφτούμε σοβαρά για κάποιες περικοπές και εξοικονομήσεις κονδυλίων για να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει Μία λεπτομέρεια θέλω να ε, δω. Ε, είχα ε, ασκήσει επίκριση ότι δεν έχουμε ένα business plan. Αν ξεκινήσουμε ένα τέτοιο εγχείρημα, πρέπει με κάθε λεπτομέρεια να έχουμε σχεδιάσει το τι θα γίνει, Όπω απαιτούμε να γίνεται και με άλλα εγχειρήματα. Απομένουν κάποια ερωτήματα που εκκρεμούν. στι guidelines, στι κατευθυντήριες γραμμέ, ανήκει για ένα νέο εγχείρημα να έχουμε σαφείς λεπτομέρειε στα κονδύλια τι θα γίνει. Και είπε ο συνάδελφος ε, ότι θα έχουμε 13 εκατομμύρια εκατομμύρια διοικητικέ δαπάνε και ότι είναι ανοιχτό λέει αυτό ε, και προ συζήτηση. Από την άλλη πλευρά έχουμε κάποιο, κάποια αριθμητικά μεγέθη, πόσα στελέχη θα προσληφθούν, δεν είναι ακριβή οι λογαριασμοί ακόμα, πόσοι θα είναι συνεργάτε ε, και ποιοι θα είναι επικεφαλεί σε, σε αυτό τον οίκο τη Ευρώπη. Αν όμω θέλουμε να λειτουργήσει αυτό ο οίκο τη Ευρώπη, πρέπει να είναι καταλεπτό σχεδιασμένα όλα αυτά και να είναι σαφεί όλε οι λεπτομέρειε. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε έτσι γενικόλογα. Δημιουργείται δυσκολία με κάτι τέτοιο. Πρέπει να υπάρχει ένα σαφέ ε, ποσό και να υπάρχει ένα business plan. Δεν μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε στα τυφλά. Έχω αμφιβολίε λοιπόν. Ακόμα και αν υπάρχουν καλοί λόγοι, καλά επιχειρήματα υπέρ του εγχειρήματο, δημιουργούνται πολλά προβλήματα όσον αφορά την κατάσταση του προπολογισμού στο Ευρωκοινοβούλιο και πρέπει πρώτα να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα και τι λεπτομέρειε και μετά να είμαστε σε θέση υπεύθυνα να τοποθετηθούμε υπέρ αυτού του εγχειρήματο. Σοσιαλδημοκρατία δημοκράτες προανήγγυλαν ότι το σύνολο των 16 εκατομμυρίων θα το εγγράψουν πάλι στο αποθεματικό διότι θέλουν να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα προτού δώσουν το τελικό πράσινο φως, το τελικό ναι υπέρ αυτού του εγχειρήματο. Πρέπει όλες οι λεπτομέρειες να αποσαφινιστούν προτού δώσουμε λοιπόν το πράσινο φω Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα εδώ πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κύριο Αντιπρόεδρο Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ και τούτου λεχθέντος ε, να πω ότι ίσως θα σας εκπλήξει αλλά είμαι ε, ε καθηγήτρια ιστορίας ε, καθηγητής ιστορίας και δεν θα πρέπει εδώ να αγνοηθεί αυτό και γνωρίζω σε σχέση με τα μαθήματα αυτά πόσα πρέπει να αναφέρονται τα θέματα της ιστορίας. Έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι οι πραγματογνώμονες θα μεριμνήσουν για τα θέματα ουσίας. Δεν θα πρέπει να έχουμε κάποιες αμφιβολίες ή να ανησυχούμε για το πώς για παράδειγμα η επανάσταση στη Γαλλία θα παρουσιάζεται. Οι ηγετικές προσωπικότητες ε, σίγουρα οι επαΐοντες θα μπορέσουν να τα παρουσιάσουν σωστά. Και γενικά βρίσκουμε ότι είναι ένα πολύ καλό, θετικό εγχείρημα, πολύ καλό σχέδιο. Θα υπάρξει θετική πρόσθετη αξία υπέρ της Ευρώπης. Πώς όμως θα υλοποιηθούν όλα αυτά πρακτικά, χειροπιαστά. Πρέπει να διασφαλίσουμε και να μεριμνήσουμε τα διοικητικά έξοδα, οι διοικητικέ δαπάνε ε, να είναι σε ένα σωστό πλαίσιο και τα κονδύλια τα οποία θα διατεθούν και αυτά να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά και να είναι ανταποδοτικό αυτό το εγχείρημα σε σχέση με τις δαπάνες και τα έσοδα. Θα πρέπει εμείς να μεριμνήσουμε στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο να ρυθμιστούν όλα αυτά. Είναι ένα μεγαλόπνο εγχείρημα σε ένα μεγαλύτερο χρονορίζοντα. Πρέπει να δεσμευτούμε και να πούμε θα δημιουργηθεί πρόσθετη αξία για την Ευρώπη από αυτό το εγχείρημα και να μεριμνήσουμε να είναι προσιτές οι να είναι βιώσιμο ας το πω έτσι αυτό το εγχείρημα σε σχέση με τις δαπάνες. Και όσον αφορά το περιεχόμενο, την ίδια την ουσία έχουμε τους πραγματογνώμονες, έχουμε τον ε, καθηγητή για παράδειγμα από την ε, ε, Φινλανδία, τον κύριο Κλίνε και τους επαΐοντες που θα μπορέσουν με τον καλύτερο τρόπο να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, καλύτερα από ό,τι μπορούμε εμείς ως Ευρωβουλευτές να δώσουμε απαντήσεις. Και πριν από τις εκλογές Σίγουρα καλό θα ήταν να λέγαμε ότι γνωρίζουμε καλύτερα εμείς αυτά τα πράγματα από, από άλλοι. Είναι δική μας δουλειά το εγχείρημα αυτό να προαχθεί και εμείς να μεριμνήσουμε ώστε οι τεχνικές λεπτομέρειες να μπορέσουν να διευθετηθούν και τα πράγματα να πάνε καλά. Ήθελα με τα λόγια αυτά, με την παρέμβασή μου να ενθαρρύνω και να υποστηρίξω, να εκφράσω την υποστήριξή μου για αυτό το εγχείρημα. Και η ομάδα μου το υποστηρίζει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Τρεις έχουν ζητήσει ακόμα τον λόγο και κλείνω τον κατάλογο αγορητών. Μπόρις, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας κάποια πράγματα έχουν αλλάξει Έχουμε πλέον μια ενιαία ιδιότητα Ευρωπαίου πολίτη, έχουμε κοινέ πρωτοβουλίες όπως την πρωτοβουλία των πολιτών και έφτασε η στιγμή να πούμε ότι η ιστορία της Ευρώπης θα πρέπει να ξαναβρει τη θέση που της αξίζει. Στην Ευρώπη μπορούμε να βρούμε πάρα πολύ καλά παραδείγματα για τον πολιτισμό, την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά ή την φιλοσοφία και ό,τι άσχημο επίσης μπορούμε να το βρούμε στην Ευρώπη που έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να δώσουμε στις επερχόμενες γενιές την δυνατότητα να γνωρίσουν το σύνολο της Ευρώπης και το σύνολο των χωρών της, της Ευρώπης και την ιστορία τους. Μέχρι τώρα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τουλάχιστον το ε, μέγεθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ενήμεροι για την κατάσταση. Πρέπει οι πολιτικές ομάδες να γνωρίζουν επίσης το τι μπορούμε να δημιουργήσουμε ή τι έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα και πρέπει να υπάρξει από πλευράς όλων των πολιτικών ομάδων ε, μια αποδοχή του συγκεκριμένου προγράμματος. Σχετικά τώρα με τη χρηματοδότηση θα πρέπει τα πράγματα να τα κάνουμε σωστά. Θα πρέπει εμείς να καταστήσουμε το μουσείο αυτό ελκυστικό στη μορφή του, να χρησιμοποιήσουμε τα παραδείγματα των σύγχρονων μουσείων. Υπάρχει το Μουσείο του Τρόμου στην Βουδαπέστη, να ένα παράδειγμα ενός μουσείου με μεγάλο ενδιαφέρον. Το Μουσείο του Τρόμου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται το Μουσείο του Τρόμου σε ετήσια βάση. Θα πρέπει λοιπόν και το περιεχόμενο αλλά και τη μορφή να φροντίσουμε. Εφόσον λοιπόν υπάρξει μια αποδοχή του συγκεκριμένου προγράμματος τότε θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε επίπεδο χρηματοδότησης. Δεν θα πρέπει να εμείνουμε στο θέμα της ετήσιας χρηματοδότησης. Ξέρω ότι η, πρόταση είναι μια δύσκολη, περίπλοκη πρόταση, αλλά εν πάση περιπτώσει εφόσον μπορούμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, πρέπει ε, να το, αποφασίσουμε για τα επόμενα 5 ή 7 χρόνια. Ευχαριστώ, δεν θα επανέλθω στο περιεχόμενο του σχεδίου αυτού και σε τεχνικό και σε πολιτιστικό επίπεδο. Αλλά στην παρουσίαση όλων όσων πήραν το λόγο μέχρι τώρα, τίθεται το οικονομικό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει συγκεκριμένες βαρύτατες οικονομικές επιβαρύνσεις. Ξέρουμε επίσης ε, ε, την ε, δημοσιονομική λιτότητα μέσα στην οποία ζούμε θα ασκηθεί κριτική στην απόφασή μας. Ε, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τα δημοσιονομικά και να επανέλθω σε κάτι το οποίο έχει σημασία όταν συζητάμε τόσο σημαντικά θέματα. Πρέπει να λειτουργήσουμε παιδαγωγικά. Πρέπει να εξηγήσουμε και τη σημασία που έχει από τη μία η οικονομική πλευρά και από την άλλη το περιεχόμενο αυτής της πρωτοβουλίας. Ε, έχει γίνει μια συζήτηση και εφόσον συνεχιστεί θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα τα επιχειρήματά μας σχετικά με τη σημασία που έχει το πρόγραμμα αυτό. Θα πρέπει ένα τέτοιο πρόγραμμα να συνοδεύεται από ένα παιδαγωγικό σχέδιο υπόβαθρο. Πρέπει να είναι ένα μουσείο και των παιδιών και των νέων απέναντι σε όλους τους συμμετέχοντες και είναι πολύ θα έλεγα έτσι ώστε να καλύψουμε όλες τις ιστολικές και παιδαγωγικές πλευρές. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Μαρτίνες Μαρτίνες Μαρτίνες για την παρουσίασή του. Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να πω ότι η ιστορία δεν είναι απλά ένα σύνολο εθνικών ιστοριών. Υπάρχουν σημαντικά θέματα τα οποία τίθενται και σε επίπεδο πολιτιστικό. Και γι' αυτό ακριβώς αυτός ο οίκος της ευρωπαϊκής ιστορίας είναι κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη. Ανήκω στην ομάδα εργασίας για τη συμφιλίωση η ιστορία αυτή η ομάδα εργασίας έχει ε, τους ίδιους στόχους. Θέλουμε να αναφερθούμε στην κοινή ε, θα έλεγα καταγωγή μας στις κοινέ εξελίξεις και στην συνειδητοποίηση ε, από κοινού των προβλημάτων πάντα θέτοντας φυσικά, υπογραμμίζοντας το μέλλον, γιατί εκεί πρέπει να είμαστε προς τα εκεί. Μάλιστα, εντάξει, παρακαλώ Μιγέλ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο γίνεται πιο σύντομα. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Πρέπει να σας πω ότι κάποια στιγμή με την κυρία Τρούπελ υπό τη δικιά της ιδιότητα ε, συζητήσαμε και θεωρήσαμε πολύ χρήσιμη την συμμετοχή της και επιβεβαιώνω ότι είναι ε, μία βουλευτής η οποία έχει δημοσίευση άρθρο, το οποίο το έχω βάλει και εγώ στους φακέλους μου για να το δείχνω, για να ξέρει ο κόσμος ότι το στηρίζει. Όλα τα ερωτήματά σας είναι απόλυτα ουτιολογημένα και πρέπει να σας δώσω μια απάντηση. Στον κύριο Καβαντά, πρώτα απ' όλα. Καταλαβαίνετε κύριε Καβαντά, μερικές φορές ε, με συγκινείτε. Ειλικρινά κύριε Καβαντά, αυτά που είπατε με τόση ειλικρίνεια, τι Όλα αυτά πρέπει να τα μάθουν και οι συνάδελφοι. Εσείς είσαστε άνθρωπος της επικοινωνίας και ελπίζω πραγματικά ότι μπορούμε να βασιστούμε σε εσά για να μεταφέρετε το μήνυμα αυτό που μπορείτε να το μεταφέρετε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον. Αναφερθήκατε στο ρόλο του Πέτερινγκ. Θέλω να το πω και εδώ, γιατί το έχω πει και στο Προεδρείο, ότι μερικές φορές δεν χαίρονται όλοι για αυτά που λέω. Ο Hans Gert Πέτερινγκ παίζει έναν αξιοθαύμαστο ρόλο. είναι κάποιο που χαίρει ιδιαίτερου σεβασμού και στη χώρα του και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη διεθνή σκηνή. Ασχολείται με μια δουλειά που τον ενθουσιάζει, όπως και εμένα. Πρόεδρος του Ιδρύματος Κόντρα Ταντενάουερ, ξέρουμε πολύ καλά όλοι τι κάνει στον κόσμο το Ίδρυμα αυτό. Άρα λοιπόν ο ίδιος δεν το έχει ανάγκη. Αν ε, το κάνει και θέλει το σχέδιο αυτό, είναι γιατί πραγματικά τον παθιάζει, τον ενθουσιάζει, το θέλει. Και είναι εξωθαύμαστος. Και το λέω αυτό σε ανθρώπους που δεν θεωρούν ότι ο Πέτερινγκ είναι ε, στο πλευρό τους ιδεολογικά ή από πλευράς ε, θρησκείας Κοιτάξτε, βλέπετε οι χριστιανοί θεωρούν ότι έχουν την αιώνια ζωή. Εμείς βλέπουμε τα πράγματα πιο μεσοπρόθεσμα. Μας ενδιαφέρει τι θα γίνει πιο σύντομα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, θα έλεγα ότι ζηλεύω. Ζηλεύω, κύριε Καβαντά. Ο Ρωμάνο ε, φίλος που ήταν εδώ αναφέρθηκε στις αξίε Και, κύριε Χάνεμπολ, εσεί ρωτάτε μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Κύριε Χόνεμπολ, πρέπει να σας πω. Ανάμεσα στα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε υπάρχουν εμπόδια διαφορετικών ειδών. Υπάρχουν άνθρωποι που από την αρχή είναι κατά του σχεδίου αυτό, γιατί είναι κατά της Ευρώπης και το έχουμε δει αυτό σε ορισμένες ομάδες, όπου συμμετέχουν διάφοροι από ορισμένε χώρες. Υπάρχει εχθρότητα απέναντι στο σχέδιο αυτό που έχει να κάνει με το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι πρέπει να χάνουμε ούτε ένα λεπτό συζητώντας μαζί τους. Είναι κατά και στο κάτω-κάτω και συνεπείς με την άρνησή τους αυτή. Είναι συνεπείς με τις ιδέες τους και αναφέρουν επιχειρήματα και κινητοποιούν και τα μέσα ενημέρωση μερικέ φορέ με τα επιχειρήματά του. Γιατί βέβαια είναι πιο εύκολο να κινητοποιήσει κανεί προ αυτή την κατεύθυνση τα μέσα ενημέρωση παρά προ την άλλη που λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Αναφερθήκατε στην ε, διαδραστικότητα και στο περιεχόμενο του σχεδίου. Όσον αφορά το σχέδιο, πρέπει να το συζητήσετε με τη διευθύντρια του μουσείου. Εκείνη θα σας παρουσιάσει το περιεχόμενο. Τώρα θα σας μεταφέρω μια προσωπική άποψη. Η μόνιμη έκθεση θα πρέπει να είναι πολιτικά ουδέτερη, χωρίς να στρεβλώνει βέβαια τις αρχές, αλλά πολιτικά και κομματικά ουδέτερη. Ε, δεν σημαίνει ότι θα βασιστούμε σε αυτούς που είναι κατά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο πλουραλισμός που εκπροσωπούμε εδώ θα προβληθεί πιο πολύ στην ε, προσωρινής διάρκειας ε, έκθεση. Ας πούμε μπορούμε να κάνουμε μια έκθεση για τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή στην ιστορία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ή μπορούμε να μιλήσουμε για τον χριστιανισμό στην Ευρώπη σε αυτές τις περιοδικές εκθέσεις. Και εδώ πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον για να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους να παρουσιάσουν βέβαια μέσα σε ένα ε, συγκεκριμένο πλαίσιο που θα δείχνει σεβασμό προς όλους να παρουσιάσει τις απόψεις τους. Οι πράσινοι ας πούμε θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να κάνουν μια έκθεση για παράδειγμα, για την πυρηνική ενέργεια. Γιατί όχι, στην Ευρώπη. Γιατί όχι. Και εγώ είμαι πρόθυμος για όλα αυτά στις μη μόνιμες εκθέσεις, στις περιοδικές εκθέσεις δηλαδή. Και εκεί θα υπάρχει διάδραση με μουσεία ή με πολιτιστικά κέντρα, και, έχουμε και πανεπιστήμια, γιατί έχουμε ήδη πολλά πανεπιστήμια που ενδιαφέρονται. Βλέπετε υπάρχει το διαδίκτυο που δίνει νέε δυνατότητες και είναι ενημερωμένοι μερικές φορές περισσότερο από ορισμένους εδώ μέσα και θέλουν να παρακολουθούν τι γίνεται με αυτόν τον οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Τώρα για αυτό που είπε η κυρία Τρούπελ. Εκφράζω κάθε σεβασμό και θαυμασμό προς το πρόσωπό της. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει. Έχει την ευθύνη του προπολογισμού, οπότε έχει ακόμα περισσότερα ε, προβλήματα, γιατί συγχρόνως υποστηρίζει και το σχέδιο. Αυτό το καταλαβαίνω, την καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Όσοι είναι στην Επιτροπή Προπολογισμού, δεν λέω, σέβονται το σχέδιο και όσοι είναι στην Επιτροπή Πολιτισμού συγχρόνως πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και τις ανησυχίες τις δημοσιονομικές. Αναφερθήκατε σε ένα business plan. Εκπονείται και θα είναι έτοιμο μέσα σε μερικές μέρες ή εβδομάδες. Για να είμαι όμως απόλυτα ειλικρινής με όλους σας. Προσωπικά δεν έχω συμμετάσχει σε αυτό. Βλέπετε είναι αλήθεια ότι σε τέτοιου είδου σχέδια μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο για την πολιτική πλευρά να πάει και να πει ποιο είναι το business plan. Δεν λέω το χρειαζόμαστε, αλλά δεν μπορεί να το κάνω εγώ αυτό, ούτε ο κύριος Καβαντά. Άλλοι θα το κάνουν που γνωρίζουν καλύτερα αυτά τα πράγματα. Ακόμα και όρος business plan. Για μένα, τι να σας πω. Δεν ξέρω, εγώ ούτε plan ούτε business είμαι. Οπότε, αλλά θα γίνει, θα γίνει. Υπάρχει κάτι που θέλω να καταλάβετε, κυρίως η κυρία Τρούπελ. Έχω πιέσει πάρα πολύ για να μην ε, ακούμε υπερβολές. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολο να βγάλει κανείς από το κεφάλι του ποσά και να λέει αυτό θα στοιχήσει 7 εκατομμύρια. Γιατί είτε πεις ότι θα στοιχήσει 7 εκατομμύρια, είτε πεις ότι θα στοιχήσει 27 εκατομμύρια, το ίδιο σου στοιχίζει. Εύκολο είναι να πεις θα στοιχήσει 15 εκατομμύρια, ενώ ξέρουμε ότι θα στοιχήσει 60. Δεν έχει σημασία. Πάλι 7 θα πει ο άλλος, γιατί είναι πιο εύκολο να περάσει το 7 παρά κάτι παραπάνω. Ε, όχι λοιπόν. Τα ποσά που βάζουμε είναι λογικά ποσά. Θα μπορέσουμε να τα τηρήσουμε. Και τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. 60 εκατομμύρια. Είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό. Ε, ναι, είναι. Μεγάλο. Τι σημαίνει στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ποιος είναι ο προπολογισμό των γραφείων που ανοίγουμε του Κοινοβουλίου σε κάθε πρωτεύουσα και μερικές φορές όχι μόνο στις πρωτεύουσες αλλά και σε δύο και σε τρεις πόλεις στην ίδια χώρα. Θέλουμε να δώσουμε λεφτά για θέματα επικοινωνίας. Εντάξει, να τα δώσουμε, αλλά να δούμε πόσα είναι. 6-600. Εδώ μιλάμε για 60 εκατομμύρια και λέτε «Α, πολλά». Αλλά η εμπειρία μου από τον πολιτισμό είναι ότι όλα είναι υπερβολικά ακριβά και δεν υπάρχει ποτέ χρόνος, γιατί πάντα βρίσκουμε άλλες προτεραιότητες. Πάντα υπάρχει κάποια άλλα προτεραιότητα που πιέζει περισσότερο. Αν όμως δεν θεωρήσουμε τις αρχές μας και τις αξίες μας ως προτεραιότητα, ως την προτεραιότητα, ε, τότε ας βγούμε από το παιχνίδι. Και υπάρχει κάτι που με κνευρίζει μερικές φορές. Αυτό είναι το θέμα των μέσων ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης έτσι κι αλλιώς θα ασχοληθούν και ασχολούνται καθημερινά με τα πάντα. Έρχονται λοιπόν και ψάχνουν αν κερδίζουμε υπερβολικά πολλά ποσά αναφέρουν που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Το κάνουν. Δεν μπορούμε εμείς να δουλεύουμε όντας όμοιροι των μέσων ενημέρωσης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το τι λένε, σύμφωνοι, αλλά πρέπει και να τολμήσουμε. Γιατί αλλιώς εγκαταλείπουμε τις δικτατορίες που πολλοί από μας γνώρισαν για να μπούμε σε ενός νέου είδους δικτατορία που θα είναι τα μέσα ενημέρωσης. Όσοι έχουμε περάσει τη μισή μας ζωή να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία του τύπου, βέβαια αυτή η κατάσταση είναι παράδοξη και θέλουμε να την αποφύγουμε. Θέλω να πω και δύο λόγια στον κύριο Μπόρις τώρα. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Οι Πολωνοί έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο σχέδιο αυτό και χαίρομαι πολύ ένας από αυτούς που έπαιξε ένα ρόλο κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η Μαρία Σμιτ, που είναι η πρόεδρος ε, του Μουσείου της Βουδαπέστης, στο οποίο αναφερθήκατε. Είναι στην ίδια γραμμή, λοιπόν, με αυτά που κάνουμε. Και ακόμα και αν μερικές φορές έχω την αίσθηση, ειλικρινά σας το λέω, ότι δεν έχουμε δουλέψει τόσο επαγγελματικά επειδή βασιζόμαστε σε αξίες, σε ιδέες, μπαίνουμε με ενθουσιασμό στο σχέδιο και ίσως μερικές φορές να παρατηρείτε έλλειψη επιστημονικότητας ή επαγγελματισμού, πράγμα το οποίο οδηγεί σε προβλήματα οικονομικά. Από την άλλη χαίρομαι που αναφερθήκατε σε αυτό το μουσείο, γιατί η Μαρία ήταν το πρόσωπο κλειδί στην επιλογή του προσωπικού. Έχετε δίκιο λοιπόν. Και κάτι τελευταίο που ξέχασα και με ρωτήσατε, το σχολιάσατε. Ένα από τα πράγματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι συνάδελφοι έχει να κάνει με αυτό που είπε και η Μαρία Τερές. Έχουμε το κέντρο επισκεπτών, λένε μερικοί. Ε, ας το κάνουμε στο κέντρο επισκεπτών, γιατί θέλουμε κάτι άλλο για να μην συζητήσουμε τώρα πόσο στήξε το κέντρο επισκεπτών και πόσο θα κοστίσει ακόμα. Όμω εμεί θέλουμε να φτιάξουμε ακριβώ αυτό το τρίγωνο. Δηλαδή κέντρο επισκεπτών, μουσείο, ημικύκλιο. Το μουσείο αυτό έχει κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Όταν ανήκει κανείς ένα μουσείο, η ερώτηση είναι ποιος θα μπει στο μουσείο αυτό. Εμείς μόλις θα ανοίξουμε ένα εκατομμύριο θα έρθουν αμέσως. Γιατί ένα εκατομμύριο άνθρωποι έρχονται και επισκέπτονται τα κτίρια μας στις Βρυξέλλες. Ομάδες επισκεπτών επίσης που έρχονται από μόνες τους, όχι μόνο αυτές που προσκαλούν τα πολιτικά, οι πολιτικές ομάδες, θα είναι λοιπόν το μοναδικό μουσείο στον κόσμο όπου οι άνθρωποι δεν θα έρχονται τόσο ατομικά, θα έρθουν ατομικά βέβαια, έρχονται σε ομάδες. Και ορισμένοι μας είπαν, το μουσείο αυτό πρέπει να το κάνουμε μια ελκυστική πλατφόρμα για τουρίστες και για ανθρώπους που επισκέπτονται τις Βρυξέλλες. Οι άνθρωποι λοιπόν υπάρχουν, οι επισκέπτες υπάρχουν του μουσείου αυτού. Και γι' αυτό που λέει ο κύριος Βέρτ, Το αντιλαμβανόμαστε, το γνωρίζουμε. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε τώρα, και με αυτό θα τελειώσω, είναι τι μηχανισμούς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εφεξής ώστε να βελτιώσουμε την τυπική, την νομική πτυχή της δουλειάς μας. Γιατί από την αρχή, μην τα πείτε παραπέρα, αλλά από την αρχή πρέπει να σας πω ότι βρέθηκα σε κάπως δύσκολη θέση γιατί είχα την αίσθηση ότι έλειπε η κοινοβουλευτική δομή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων κλπ. Και αυτοί που μου είπαν, κοίτα καλύτερα θα πάει έτσι, γιατί αλλιώς αν θέλουμε να ακολουθήσουμε την παραδοσιακή οδό λήψης αποφάσεων, η μία επιτροπή, η άλλη επιτροπή κτλ, δεν θα προχωρήσουμε. Και γιατί ο Πέτεριν και εγώ κατά κάποιο τρόπο βιολογικά έχουμε δεσμευθεί πριν από τον Ιούνιο του 2014 να έχει ξεκινήσει το μουσείο. Αν μπούμε σε καινούργια κοινοβουλευτική θητεία με 50-40% ανανέωση των μελών θα πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν. Είναι όπως η οικοδόμηση της Ευρώπης. Γυρνάμε γύρω γύρω γύρω γύρω και στο μεταξύ οι υπόλοιποι παγκόσμιοι εταίροι προχωράνε πιο γρήγορα από εμά. Ε, λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να βρούμε ένα μηχανισμό. Η Επιτροπή Πολιτισμού σίγουρα θα παίξει ρόλο κλειδί για να εξασφαλίσουμε την κοινοβουλευτική συμμετοχή, τη δημοκρατική συμμετοχή στο σχέδιο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα καλά σας λόγια και την κατανόησή σας. Σε ευχαριστούμε πολύ Μιγέλ. Λοιπόν, αν τα είχαμε κάνει αυτά έτσι όπως κανονικά γίνονται κάποια πράγματα, τότε δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Και επειδή το ξέραμε αυτό, δεν τα κάναμε τα πράγματα έτσι. Αν είχαμε κάνει διαφορετικά με το Lux Prize, το βραβείο Lux ε, για τον κινηματογράφο, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Πρέπει να βοηθάει κανείς οι ιδέες να μπορούν να υλοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Φυσικά είμαστε ένα νομοθετικό όργανο. Δεν μπορούν όμως όλα να γίνονται νομοθετικά. Ας είμαστε πιο δημιουργικοί και καινοτόμοι. Πράγματα που έχουν αξία και είναι αξιόλογα για μας να τα ζωντανεύουμε και να τα συνοδεύουμε κοινοβουλευτικά. Πρέπει να συμφωνήσουμε για αυτά με την Επιτροπή Προϋπολογισμών βέβαια για τα κονδύλια, αλλά θα τα καταφέρουμε σίγουρα. Και για τα business plans δεν είναι μόνο αυτά, αλλά έχουμε ανθρώπους που συνεργάζονται για αυτή την κατεύθυνση. Χαίρομαι ότι έχουμε αυτή την κυρία, θα την προσκαλέσουμε εδώ να μας πει για το περιεχόμενο όλων αυτών και την ουσία τους. Σήμερα ευχαριστώ για την παρουσία λόγια σας, για το μεγάλο ενθουσιασμό και τη ζέση, την φλόγα σας. Είμαστε όλοι υπέρ, το βλέπετε αυτό. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει από ανθρώπους όπως σαν την Helga Trupper που είναι υπέρ, αλλά που πρέπει να προετοιμάσουν και τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για να υποστηριχθεί το εγχείρημα, να λειτουργήσουν σωστά. Και η Κωνσταντσε είναι τέλεια και έχετε πολύ καλούς ανθρώπους που θα συνεργαστούν κάθε επιτυχία και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ αγαπητέ Μιγέλ. Γεια. Για το βιολογικό ζήτημα, συμφωνώ και εγώ μαζί σας. So, coming to the next... Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο σημείο. Το σύστημα Ευρωπαϊκών Σχολείων. Ο κύριος Καβαντά, παρακαλώ, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, Présidente. Euh, ε, Ευχαριστώ συναδελφοί. Το θέμα αυτό απασχολεί πολύ κόσμο στα ευρωπαϊκά όργανα και γι' αυτό πρέπει να γίνει μια προπαρασκευαστική προσπάθεια να συναντηθούμε με όλους τους εμπλεκομένους. Για να σας παρουσιάσω μια έκθεση η οποία να είναι αξιόπιστη προσπαθούμε να συλλέξουμε τις περισσότερες δυνατές γνώμες και να συναντηθούμε με τους πρωταγωνιστές από τη Γενική Γραμματέα των Σχολείων με την εκπρόσωπο των ε, συλλόγων γονέων, τον εκπρόσωπο των καθηγητών και ε, όλους όσους εμπλέκονται εν πάση περιπτώσει. Επί τη βάση όλων αυτών Πιστεύουμε ότι για να μπορέσουν τα σχολεία αυτά να ζουν και να εξελίσσονται θα πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση επί τη βάση της λογικής της επένδυσης για το μέλλον των νέων Ευρωπαίων και όχι μόνο επί τη βάση μόνον του κόστους. Να θυμίσω ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία δημιουργήθηκαν για να υπάρξουν κάποιες δυνατότητες για τους εργαζομένους στα ευρωπαϊκά όργανα να δώσουν ένα πλαίσιο πολιτισμικό και εκπαιδευτικό στη γλώσσα των παιδιών και να μπορέσουν αν θέλουν να επιστρέψουν στην ε, χώρα τους χωρίς να νιώθουν απόμακρα. Το παιδαγωγικό πρόγραμμα των σχολείων των Ευρωπαϊκών είναι πολύ φιλόδοξο, απαιτητικό και αυστηρό. Κοινός παρανομαστής είναι η προετοιμασία ενός ευρωπαϊκού μπακαλωρεά που βασίζεται σε ένα κοινό σχολικό πρόγραμμα στη μητρική τους γλώσσα. Η ε, δευτεροβάθμια εκπαίδευση προετοιμάζει για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση σωστά και η απόκτηση αυτού του ευρωπαϊκού μπακαλωρεά δίνει κατά προτεραιότητα ένταξη σε πανεπιστήμια γιατί εγγυάται δύο ή τρεις γλώσσες στα πανεπιστήμια των χωρών της Ένωσης. Η διδασκαλία των γλωσσών φυσικά ευνοείται, η γενική διδασκαλία ε, χορηγείται σε εισαγωγικά στη μητρική γλώσσα του μαθητή, η μαθητεία μιας πρώτης ξένης γλώσσας υποχρεωτική από την πρώτη δημοτικού ανάμεσα στις τρεις βασικές λεγόμενες γλώσσες, τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. Σε αυτές τις γλώσσες λοιπόν μετά από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάσκονται τα μαθηματικά και οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Περνάμε δηλαδή από την εκμάθηση των γλωσσών σε ένα ανώτερο επίπεδο. Η βασική αρχή μιας πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης επί της οποίας βασίζεται η ευρωπαϊκή, τα ευρωπαϊκά σχολεία αναπτύσσει τις ευρωπαϊκές αξίες ε, με βάση τις αρχές της αμοιβαίας κατανόησης, του αμοιβαίου σεβασμού και της ανοχής. 50 χρόνια βέβαια μετά από τη δημιουργία του πρώτου σχολείου, η έννοια του σχολείου αυτού θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες θα πρέπει να παραμείνουν πρότυπο έμπνευση για τα εθνικά σχολικά συστήματα που αξιοποιεί την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη και να ευνοεί την κινητικότητα και την εκπαίδευση. Υπάρχουν δύο βασικές δυσκολίες οι οποίες έχουν αρχίσει να γίνονται ιδιαίτερα ανησυχητικέ για, αυτά τα, για αυτά τα σχολεία. Το πρώτο είναι δημοσιονομικό το πρόβλημα γιατί παρά όλα τα πλεονεκτήματα του συστήματος από την, ε, με βάση τις αρχές λειτουργίες τους ε, είναι ε, κάτι το οποίο κοστίζει. Η διδασκαλία στη μητρική γλώσσα έχει γίνει περίπλοκη μετά από τη διεύρυνση γιατί υπάρχουν πολλές γλώσσες χώρες και προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη αποσπούν εκπαιδευτικούς τους για τη διασφάλιση της διδασκαλίας στη μητρική γλώσσα των μαθητών. Αλλά σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης όπου κάθε χώρα προσπαθεί να κάνει οικονομία τα κράτη τα οποία πρέπει να στείλουν διδάσκοντες όπως η Αγγλία και η Γαλλία δέχονται όλο και λιγότερο να αποσπούν καθηγητές. Να λοιπόν ένα βασικό θέμα. Η πίεση λοιπόν επί του κοινοτικού προϋπολογισμού αυξάνεται γιατί για τους ε, ε, καθηγητές που αποσπώνται και που ε, αμείβονται σύμφωνα με τους μισθούς των χωρών τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπληρώνει το εισόδημά τους έτσι ώστε όλοι να έχουν ένα ταυτόσιμο μισθό. Είναι ενδιαφέρον βέβαια το σύστημα αυτό εκεί όπου οι μισθοί των εκπαιδευτικών είναι χαμηλοί αλλά είναι κάτι που επιβαρύνει πολύ τον προϋπολογισμό της κοινότητας. Λόγω ακριβώς και της έλλειψης αποσπόμενων εκπαιδευτικών, ένας όλο ένα μεγαλύτερος αριθμός καθηγητών προσλαμβάνονται άμεσα από τα σχολεία και πληρώνονται επί τη βάση του κοινοτικού τιμολογίου, θα έλεγα κάτι το οποίο χειροτερεύει και αυξάνει ε, το οικονομικό κόστος. θα πρέπει να ελεγχθούν οι δαπάνες και θα πρέπει να υπάρξουν και νέοι πόροι έτσι ώστε να υπάρξει μια οικονομική ισορροπία. Η τάση τα δύο τελευταία χρόνια είναι να δίδουμε έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό στα ευρωπαϊκά σχολεία, 160 εκατομμύρια ευρώ το 2010, 164 το 11 και το 12, για να περιορίσουμε το κόστος με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα διαχείρισης για τα όργανα αυτά, για τα σχολεία και σε επίπεδο επιμελητιακό και σε επίπεδο παιδαγωγικό. Το θέμα είναι πώς θα διευκολύνουμε την κινητικότητα των εργαζομένων και πώς θα φέρουμε σε επαφή τα σχολεία αυτά με τα σχολεία των κρατών μελών. Θα πρέπει να εξελιχθεί το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων λοιπόν και να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε σχολεία τύπου 2 και θα σας πω τι σημαίνει αυτό αργότερα δηλαδή σχολεία τα οποία μέσω ακριβώς μιας πιστοποίησης να υποδέχονται όχι μόνο τα παιδιά των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συμβασιούχων, αλλά και τα παιδιά των ανθρώπων που δεν είναι υπάλληλοι, εργάζονται στον ιδιωτικό χώρο και ζουν μακριά από τη χώρα τους και έχουν ανάγκη τα παιδιά τους να παίρνουν ε, ε, ευρωπαϊκή παιδεία. Όλοι ε, θέλουν οι ενδιαφερόμενοι μια τέτοια λύση. Είναι μια λύση, ένα βήμα προς μια ευρωπαϊκή πραγματικά διδασκαλία ανοιχτή σε πολύ περισσότερους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μια μεγαλύτερη αυτονομία στα σχολεία στα πλαίσια της σύμβασης που τους επιτρέπει σε ένα μεγάλο βαθμό να καθορίζουν τα ίδια τους στόχους τους και να τους δίνει ακριβώς τα μέσα για να πετύχουν τους στόχους αυτούς. Δεν θα διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των σχολείων τύπου 2, που είναι μικρά συνήθως σχολεία, παρά μόνο αν προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα μειώσουμε το κόστος και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αύξησης των ιδίων πόρων των σχολείων αυτών, τα δίδακτρα τα οποία πληρώνουν οι γονείς ε, και ε, τον, οι οποίοι δεν είναι υπάλληλοι φυσικά των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Ενώ ζητάμε από όλους τους πολίτες των κρατών μελών οικονομικές δραστικές ε, ε, παρεμβάσεις σε επίπεδο και θυσίες, σε επίπεδο αμοιβών, είναι πολύ δύσκολο η κατάσταση αυτή να μην αντικατοπτριστεί στη διαχείριση των ευρωπαϊκών σχολείων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι σε όλα τα κράτη-μέλη η παιδεία είναι δωρεάν και οι υπάλληλοι των ε, κοινοτικών οργάνων δεν έχουν άλλες δυνατότητες από το να στείλουν εκεί τα παιδιά τους εάν θέλουν τα παιδιά τους ε, να πάρουν μια σωστή παιδεία στη γλώσσα τους. Συνεπώς δεν είναι πολυτέλεια τα ευρωπαϊκά σχολεία, δεν είναι ένα δεδομένο και εκτιμένο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ε, να χρησιμοποιήσουμε και θα πρέπει όμως να το διασφαλίσουμε με νέα μέτρα και όχι εις βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης. Το μοντέλο το πρότυπο τύπου 2 ή και τύπου 3 δηλαδή σχολεία τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν μετά από πρωτοβουλία των κρατών μελών και σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη θα χορηγούν ένα ευρωπαϊκό μπακαλωρεά. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να ενθαρρύνουμε γιατί ήδη υπάρχουν βήματα προόδου ε, πολύ σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή. Η δεύτερη ανησυχία και θα τελειώσω με αυτή προέρχεται από την πρώτη. Είναι το θέμα των προσλήψεων το βασικό θέμα για την επιβίωση του συστήματος είναι πράγματι η, η μέθοδος των αποσπάσεων από διάφορα κράτη-μέλη εκπαιδευτικών. Θα πρέπει να επιθυμίσουμε λοιπόν στα κράτη-μέλη που δεν φέρουν εις πέρα στις υποχρεώσεις τους την δέσμευσή τους έτσι ώστε το ταχύτερο δυνατόν να θέσουν στη διάθεση των σχολείων τις ποσοστώσεις των αποσπόμενων εκπαιδευτικών που απαιτούνται και έχουν συμφωνηθεί Συνεπώς θέλω το προσχέδιό μου να είναι συγκεκριμένο και χρήσιμο για να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν μέσα σε ένα νέο πνεύμα τα σχολεία αυτά. Είναι ευαίσθητο το θέμα, είναι περίπλοκο το θέμα, αφορά τα παιδιά μας. Είναι κάτι το οποίο θα εξυπηρετήσει την εκπαίδευση με μια ευρωπαϊκή προοπτική. Είναι ένα πείραμα αν θέλετε το οποίο σε ευρωπαϊκό πολιτιστικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και δείχνει ακριβώς μια υποδειγματική πορεία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πιστεύω ότι με το σύνολο των σκιωδών ε, εισηγητών και με όλους τους ενδιαφερομένους θα καταλήξουμε σε μια έκθεση η οποία θα είναι καρπός της ανταλλαγής ε, απόψεων. Ο απολογισμός της λειτουργίας των ευρωπαϊκών σχολείων είναι ξεκάθαρα θετικός και νομίζω ότι η έκθεση αυτή δίνει τις δυνατότητες να δημιουργηθεί ένα νέο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα που δεν υπάρχει εκτός αυτών των σχολείων. Θα πρέπει λοιπόν με κάθε δύναμη που έχουμε να ζητήσουμε την πολιτική στήριξη των κρατών μελών και να πείσουμε τα κράτη-μέλη αυτά όχι μόνο να διατηρήσουν το σύστημα αλλά να βοηθήσουν την ανάπτυξη αυτού του πρότυπου και μοναδικού συστήματος και στις δικές τους χώρες. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την πολιτιστική ταυτότητα της εκπαίδευσης, θα πρέπει να είναι οι καθηγητές από τις χώρες στις οποίες, στον οποίο τη γλώσσα διδάσκονται τα μαθήματα, και θα πρέπει να στηρίξουμε το Ευρωπαϊκό Μπακαλωρεά που είναι υψηλής ποιότητας και να διασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη αυτονομία των ευρωπαϊκών σχολείων με οικονομικά μέσα τα οποία θα τα διαχειριστούν σωστά για να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους. Θυμάμαι και δύο άλλες εκθέσεις που είχαμε για τα ευρωπαϊκά σχολεία που ήταν α, επίμαχα θέματα από τον συνάδελφο Πέρι από τη Μεγάλη Βρετανία που είχε αναλάβει τη σύνταξη ε, εκθέσεων ιδρύθηκαν τα ευρωπαϊκά σχολεία σε μια εποχή που ήταν απλούστερα τα πράγματα να διαμορφωθούν. Τι θα κάνετε σήμερα με 23 γλώσσες με αυτά τα σχολεία. Είναι δυνατόν να λειτουργήσουν έτσι. Είναι αναγκαία καν. Δεν θα έπρεπε να μεριμνήσουμε το αποκαλούμενο Ευρωπαϊκό Απολυτήριο Γυμνασίου και αυτά που στα ευρωπαϊκά σχολεία τι τελευταίε δεκαετίε από γνώσει και από ε, ομάδε ε, ε, γνώσεων είχαν προετοιμαστεί οι δυνατότητε. Δεν θα πρέπει να χυθούν στα ε, κράτη-μέλη. Θα πρέπει σε ε, να ασχοληθούμε με αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε απλά έτσι όπω είχαμε τα πράγματα μέχρι σήμερα. Κάνω λόγο για τι 23 γλώσσε. Η ιδέα ήταν να μπορεί κανεί να μιλάει στη μητρική του γλώσσα και να σπουδάζει στη μητρική του γλώσσα. Με έξι ιδρυτικά μέλη γινόταν αυτό. Τώρα είμαστε 27 κράτη-μέλη με 23 γλώσσε. Δεν γίνονται αυτά πια. Είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα ευρωπαϊκά σχολεία με την παλαιά μορφή και τον παλαιό τρόπο. Πρώτον δεν υπάρχουν αρκετά παιδιά ώστε να υπάρχουν ομάδες ε, ε, συστάξεις ε, γλωσσικές. Δεύτερον δεν υπάρχουν επαρκείς δάσκαλοι, αρκετοί δάσκαλοι και η βούληση των κρατών να στείλουν δασκάλους είναι πολύ περιορισμένη. Παρότι πιστεύω ότι καλό θα ήταν βέβαια αν περισσότερες δασκάλες και δάσκαλοι από τις χώρες μας θα ξεκινούσαν να πάνε σε άλλες χώρες ώστε εκεί να μάθουν τι είναι η Ευρώπη διδάσκοντας στο εξωτερικό. Καλό θα ήταν αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι οι δικές μου παρατηρήσεις. Ίσως κυρία Χάνιμπαλ θέλει να πει κάτι. Παρακαλώ κυρία Χάνιμπαλ. Yes, thank you, Ευχαριστώ. Σύμφωνα απόλυτα. Ήμουνα και εγώ συγκέντρια πριν από μερικά χρόνια, οπότε έχω μια κάποια εμπειρία. Ήταν δύσκολο και γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διδάσκουμε τη μητρική γλώσσα. Από ό,τι θυμάμαι, κάποια παιδιά, για κάποια παιδιά ίσχυε το ότι οι γονείς τους δεν τους μάθαιναν καν τη μητρική γλώσσα γιατί θεωρούσαν ότι ήταν πιο χρήσιμο να μαθαίνουν κάτι άλλο. Οπότε πρέπει να δούμε τι θέλει ο κόσμος. Έχω μια ερώτηση. Θυμάμαι ότι ήταν πρόβλημα όταν εγώ έκανα την σχετική έκθεση και αυτή είναι τα αγγλικά. Οι καθηγητές, στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον, οι καθηγητές ε, προσλαμβάνονται από την τοπική αυτοδίκηση. Οπότε, αν φύγεις, δεν ξέρω αν μετά μπορείς να ξαναγυρίσεις. Δεν ξέρω στην Ιρλανδία τι γίνεται, πάντα στον Ηνωμένο Βασίλειο έτσι είναι. ίσως γι' αυτό να υπάρχει απροθυμία. Τα αγγλικά γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Η ζήτηση για τη διδασκαλία αγγλικών είναι και όλο πιο μεγάλη. Και γι' αυτό ήταν πρόβλημα η παροχή διδακτικού προσωπικού με αγγλικά μητρική γλώσσα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό, αν υπάρχουν εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση των κύριο Καβαντά. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να είναι διτό, διπλής κατεύθυνσης σύστημα. Αφενός αυτά τα οποία βλέπουμε και βιώνουμε στο, στα δικά μας θεσμικά όργανα. Τι, ποια είναι αυτά ότι λειτουργούν καλά τα πράγματα. Υπάρχουν ε, από τα εθνικά ε, Υπουργεία Παιδείας ε, οι διορισμοί τους έχουν τα πιστοποιητικά και εν μέρει είναι συγχρηματοδοτούμενη αυτή η πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει μια ιδανική λύση που να, όλα να μπορούν να λύνονται τέλεια με το μαγικό ραβδί. Πρέπει να υπάρχουν και παιδιά σε επαρκή αριθμό για τις ομάδες και τις τάξεις για να μπορούν να διδάσκονται αυτές οι γλώσσες, αυτά τα μαθήματα. Θα πρέπει όμως να κάνουμε μια αναθεώρηση. Να επισκοπήσουμε και να αναθεωρήσουμε πόσα κράτη-μέλη είναι σε θέση να υποστηρίξουν αυτά τα ευρωπαϊκά σχολεία. Διότι η κινητικότητα βρίσκεται υπό εξέλιξη. Καθοδόνα το αποκαλέσω έτσι. Και μετακινούνται οι πολίτες, αλλάζουν δουλειά, πάνε από τη μια χώρα στην άλλη. Θα έπρεπε και εμείς να προσαρμοστούμε σε αυτό και να λάβουμε υπόψη τη ζήτηση και την ανάγκη να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες στα κράτη, από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να απευθύνουμε έκκληση και στα κράτη-μέλη. Να τους πούμε αναγνωρίζουμε το πρόβλημα βέβαια, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη εμπλοκή από τα κράτη-μέλη που θα επικεντρώνονται στις μειονότητες, ώστε πραγματικά να μπορέσουν τα ευρωπαϊκά σχολεία για να προχωρήσουν σωστά. Λοιπόν, ο κύριος Καβαντά, παρακαλώ θέλετε να τοποθετηθείτε. Όχι. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Φυσικά, ξεκινάμε έτσι σιγά σιγά τις διαβουλεύσεις περισσότερο σε βάθος. Σας ευχαριστώ πάντως για την πραγματικότητα που παρουσιάζετε και εσείς και για τις ιδέες σας. Πρόεδρο, εντάξει, σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Καβαντά. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφοι. Υπαριθμό 14, το 14. Έχετε κάτι ω ένσταση κατά των αποφάσεων των συντονιστών. Όχι. 15, διάφορα. Δεν έχετε διάφορα. Υποθέτω. Εντάξει, νομίζω κάναμε σωστά τη δουλειά μα σήμερα και ολοκληρώσαμε. Επόμενη συνάντηση 11 και 12 Απριλίου. Σα εύχομαι να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο χωρίς εντάσεις και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ τους διερμηνείς.